Συνάδελφοι, καλημέρα σας. Τι προτείνω να αρχίσουμε και πάλι τις εργασίες μας από το σημείο που διακόψαμε χθες. Σε ποιο σημείο? Το 16 της ημερήσιας διάταξης. και στην εισηγήτριά μας ε, για γνωμοδότηση η Σαρία Σαγιά θα δώσω το λόγο για την έκθεσή της για δημογραφική αλλαγή και τις συνέπειές της για τη μελλοντική πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων εμείς ε, την είχαμε επεξεργαστεί αυτή την έκθεση για την ε, δημογραφία με 49 τροπολογίες που είχαν κατατεθεί και σας δίνω το λόγο κυρία μου. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι και κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Η έκθεση αυτή αφορά τις δημογραφικές αλλαγές και είναι μια σύντομη γνωμοδότηση που επικεντρώνεται κυρίως στις συνέπειες της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. Πιστεύω ότι το πνεύμα της νομοδότησης και των τροπολογιών δείχνει ότι θα πρέπει όλα τα μέτρα να συμπληρώνουν το ΑΕΠ ως στοιχείο της μελλοντικής πολιτικής. Προσπαθούμε να βρούμε ακόμα την βέλτιστη σύνταξη της γνωμοδότησης και ε, εκκρεμεί ακόμα η τελική έκδοση της έκθεσης, αλλά πιστεύω ότι μετά την τελική επεξεργασία θα έχουμε την καλύτερη δυνατόν λύση ενσωματώνοντας ε, το πνεύμα των τροπολογιών. Δύο-τρεις παρατηρήσεις έχω να κάνω. Είναι τροπολογία 31, όπου το, η παραγωγικότητα, η λέξη παραγωγικότητα, productivity, θα αντικατασταθεί με τη λέξη accessibility, προσβασιμότητα. Ε, διότι το νόημα, το νόημα της πρότασης αυτής αλλάζει τελείως αν ε, γίνει αυτή η αντικατάσταση ε, εκτός αν αναφέρουμε και τις δύο αυτές λέξεις, και την παραγωγικότητα και την προσβασιμότητα. Η τροπολογία 43 λέει ότι καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί την νομική ασφάλεια των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Και πιστεύω ότι το ε, υπόλοιπο τμήμα αυτής της τροπολογίας εμπίπτει στο πλαίσιο της ε, This opinion and I thank my της επικουρικότητας, οπότε καλό είναι να κάνουμε μια ξεχωριστή ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για να ακούσω τώρα ποιοι συνάδελφοι θα επιθυμούσαν σε αυτό το θέμα να παρέμβουν. Κύριο Σρόντερ, αλλά που εξήλθε. Σίμωρ, κύριε Σίμωρ, απούσα. Για τους κοιόδες συγγητές ε, βλέπω τον κατάλογό μου, κοιτάζω τον κατάλογό μου, δεν υπάρχουν και πολλοί. Κύριε Σαγιά, ε, θα είναι πολύ πιο εύκολο για σας έτσι, μια απλή απλή υπόθεση από ότι είναι στην πραγματικότητα. Προσπαθώ να δω τι διαθέσεις θα εμφανιστούν έτσι πρωί πρωί, αλλά... αλλά... <laughs> Δεν θα σας τσιγκλίσω για να λάβετε το λόγο. Θα περιμένω μέχρι την ψηφοφορία. Κύριε Σρέτερ, μήπως, μήπως θα θέλατε να πείτε κάτι. Όχι. Εντάξει. Κύριε Σαγιά, τι να σας πω. Συγχαρτήρια. Δεν έχω και τίποτα άλλο. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτή και για τους συναδέλφους να υπενθυμίσω κάτι ότι θα υιοθετηθεί αυτή η γνωμοδότησή, της, γνωμοδότησή σας στη συνάντησή μας στις 13 και 14 Απριλίου. Έτσι. Κύριε Σέντερ, σίγουρα δεν θέλετε να πάρετε το λόγο να πείτε κάτι για την έκθεση για την γνωμοδότηση κυρία Σεσαγιά. Εντάξει. Επιβεβαιώνουμε έτσι ότι όλα βαίνουν ομαλώς και αγαπητοί συνάδελφοι να έχουμε το διαλυματάκι για καφέ να υποφεληθείτε από αυτήν πριν ε, από αυτό το διαλυματάκι πριν να ξεκινήσουμε για την με τις τροπολογίες. Ε, συγγνώμη με τους ε, διερμηνείς που χθες υπερβήκαμε το, την, ώρα και διερκήσε περισσότερο αυτή η συνάντηση, αλλά να που σήμερα σας αφήνουμε και χωρίς δουλειά. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ στις θέσεις σας και πάλι για να ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας. Πολλές ψηφοφορίες σήμερα το πρωί. Σας προτείνω λοιπόν αμέσως να αρχίσουμε στο σημείο 17 Δεν ε, δουλεύει καλά το ρολόι σας κυρία μου. περίμενα 30. Ναι, Q30 είναι. Λοιπόν, είναι Μάρτιν Κέστλερ, Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γύρανσης, άρθρο 1, M συμβαστικό, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αρθρό 2, εισαγωγικό μέρο, εν λατινικό συμβαστικό, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 2, σημείο 1, συμβαστικό ο λατινικό, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 2, 2, το πι το λατινικό, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται και αυτό. Άρθρο 3, συγγνώμη, άρθρο 2, σημείο 3, το Q το λατινικό, συμβαστικό, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να πάμε Τώρα στην τροπολογία 130. Μετά το ορθοδιό 3 προσθέτει ένα σημείο με προφορική τροπολογία από πλευρά Κέστλερ που σας έχει δοθεί γραπτός. Παρακαλώ, 130 τροπολογία, τροποποιημένη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 2.3, συμβαστική λύση R λατινικό, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 126 του κ. Ζαμπρόφσκα υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται η πλειοψηφία καθαρά καθαρά είναι κατά το συμβαστική λύση ε, S λατινικό υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται άρθρο 3 1 2. Το ταύτο λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δαφείο 3. Το επόμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4. Το βέτο λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τι έχουμε μετά. Παραγωγός 1. Το W το υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παραγραφός 2, παραγραφός 14, την Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παραγραφός 3, το χ, το λατινικό, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παραγραφός 3, τροπολογία 150 καρνούχ, προφορική τροπολογία που έγινε δεκτή από τον εισηγητή, Τροποποιημένο λοιπόν υπέρ τη 150 κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 3, τροπολογία 19 της ε, Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 4, το ύψιλον του λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 4, τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 εισηγείται υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 5 άρθρο 5 παράγραφος 1 17 της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 παράγραφος 1 το ζήτητε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 3 τροπολογία 156 ναι, του Προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άθρο 5, συμβουλευτική τροπολογία αλφα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 3, τροπολογία 151, Τόμας Μαν υπέρ. Όχι, όχι, έχει αποσυρθεί, με συγχωρείτε. Ψηφίζουμε λοιπόν, άρθρο 6, παράγραφος 23, Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άθρο 5, 23 εισηγητού, προφορική τροπολογία μαζί, για χρήματα αφορά το θέμα, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Άρθρο 6, παράφαση 22, Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων, υπέρ κατά Δεν βλέπω καθαρά, μάλλον πολλοί απέχουν γι' αυτό. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικό. Ποιο ε, ξέχασε, λησμόνισε την κάρτα του. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Oh, πολλούς βλέπω από τις μεγάλες ομάδες. <laughs> να βγάλουμε ένα, να διαγράψουμε ένα από το ΕΛΚ και ένα από τους σοσιαλιστές. Α, ξεροκέφαλοι σοσιαλιστές, επιμένουν. Εγώ, εγώ, εγώ αποσύρω την ψήφο μου. Εντάξει τώρα, πέρας ψηφοφορίας. 8 υπέρ, 3 κατά, 33 αποχές. Εγκρίνεται πάντως. 7-24 εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158 μπακιν ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπή 25, Ζαμπρόφσκα, υπέρ. Όχι, όχι, όχι, καταπίπτει. Το 2, τροπολογία συγκριτού, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Παραγωγός 1, περιφερειακής πολιτικής. Υπέρ, κατά. Τι να σας πω, για να δούμε και πάλι, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. που μας ήρθαν και πάλι πολύ πολύ από το ΕΛΚ. Δεν γίνεται. να αποσυρθεί κάποιος έτσι φωτισμένος από το ΕΛΚ. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας, 22 υπέρ, 4 κατά, 17 οι αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφο 2 Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεν δείξατε όμως και ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε, εντάξει, ας ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά. Δύο περιφερειακής πολιτικής. Ψηφίζουμε. Πολύ, πολύ από το ΕΛΚ. Εντάξει, πέρας ψηφοφορίας. 24 υπέρ. Σαφώς, εγκρίνεται. Εκτελογική σκέψη 3. Α. Τη συμβαστική λύση υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Καρό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παραφός 3. Περιφερειακής πολιτικής υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Β συμβαστική λύση υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επιλογή 4, τροπολογία 30, κάτω, καταπίπτει αυτή. Να ψηφίσουμε την πράγμα 10 της περιφερειακής πολιτικής υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται σαφώς. Τελογική σκέψη 5 τώρα, τροπολογία συμβαστική γάμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τη σκέψη 5 τροπολογία 43 του κ. κατά καταπίπτει αυτή μετά την ε, έχουμε την 50 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 του ίδιου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 4 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. τι να σας πω τώρα. Για να δούμε και πάλι ηλεκτρονικά. Να ελέγξουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε 4 του εισηγητή. Voilà. Tout le monde a pu voter le vote clos. 32 υπέρ. 54 Λαμπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά από το 57 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9.58 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λήψη ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 4 περιφερικής, περιφερικών υποθέσεων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 τροπολογία Δεν θα τη θέλατε. Όχι, εγώ και ο συνάδελφος Μπαλτάσαρ την 60 την αποσύρουμε. Euh, alors, donc 60 est retiré. Αποσύρεται 60, 61. Κύριε Ροντζόλη, την αποσύρεται και αυτή. Όχι, όχι. Επιμένω. Ροντσόλη Μπαλτάσα υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. 61 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρα στις ψηφοφορίες, 21 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται το 11 τη 62 τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το εύτο λατινικό συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σύμφωνα με το 11 τώρα, 65 τροπολογία του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 67 κριτή υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε και αυτό ηλεκτρονικά, 67. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Alors, euh και αν ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας 20-24. Απορρίπτεται 12 το G το λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 συμβαστική λύση H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά από το 13 είμαστε στην Ι, το λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 τη λογική σκέψη 62-63, τις ψηφίζουμε και τις δύο, επειδή είναι ταυτόσιμες, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 74, εντάξει, μπορούμε να την ψηφίσουμε, κατά, εισηγητής, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 του εισηγητή, εντάξει, μπορούμε να ψηφιστεί και αυτή, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 14, δεν δουλεύει σκέψη, το G, το G, υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται παράγραφο 7 της Επιτροπής Περιχρονών Υποθέσεων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 Τόμα Μάν υπέρ Τι έγινε, 51 περνάει ή όχι. Α, αποσύρθηκε, εντάξει. Αποσύρθηκε η 51 και 75 αποσύρεται. Εντάξει, σύμφωνοι. 76. Τι είναι, καταπίπτει και η 76. Κύριε Λαμπέρ, τι σκέφτεστε εσείς γι' αυτό. Bon. Bon. Alors, le 156. 156 εγκρίνεται, άρα καταπίπτει. 14 τροπολογία 9 εισηγητή υπέρ. Μάλλον, συγγνώμη, συγγνώμη. Μόνο αν υιοθετηθεί 23. Τι έγινε με την 23. Πέρασε 23. Ναι, ψηφίζουμε. 9 εισηγητή υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Το 15. Η επόμενη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15.81 της κυρίας Λαμπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 82 τροπολογία υπέρ είναι υπέρ ο έτσι. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ε, είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Για να ελέγξουμε για την 82 ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίζουμε. Την 82. Πέρας ψηφοφορία. 18 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται. Η 84 του ιδίου. Ο κύριο Ροντζόλη τι έχει να πει. Μπαλτάσαρ και εγώ αποσύρουμε το 84. Α, λοιπόν πάμε στο 85 Λαμπέρ. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το L, η συμβαστική λύση, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τη 2016, παράγραφος 9 περιφερειακής πολιτικής, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για το σύνολο της πρώτης αυτής για την τροποποιημένη έκθεση. Να ελέγξουμε όμως ηλεκτρονικά, έτσι. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Το σύνολο της έκθεσης τροποποιημένη. Και αν ψηφίσατε, πέρας ψηφοφορίας. Όχι, εγώ δεν ψήφισα. 44 υπέρ, 0-0 τα υπόλοιπα. Ομόφωνα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν, δεν, δεν, δεν τελειώσαμε, δεν το κλείσαμε εδώ. Περιμένετε. Πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος. Ψηφίζουμε και πάλι το ίδιο. Υιοθετείτε συγχαρτήρια λοιπόν. να αλλάξουμε τα πράγματα στη μέση διάταξη. Επιτροπή προϋπολογισμών ε, είναι ανυπόμονη να ακούσει τις προτάσεις μας για το ΦΕΜ και την πορεία του. Άρα λοιπόν το 28 και 29 θα πάρουμε να εξετάσουμε αν ε, κανείς δεν είναι αντίθετος, έτσι. στην τελευταία σελίδα του καταλόγου ψηφοφορία σας, Τελευταία, τελευταία σελίδα. Δύο τελευταία σημεία. Ίσως να είναι και σε ξεχωριστό φύλλο, γιατί υπήρξε μια προφορική τροπολογία την τελευταία στιγμή. Για να μην χάνουμε καιρό. Για το 28 λοιπόν. Δεν χρειάζεται πανικό, θα τα καταφέρουμε. Στο 28 λοιπόν έχετε ένα κατάλογο ψηφοφορίας. Παναλαμβάνω. Μιλάμε για την κινητοποίηση του ΦΕΜ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής, για την Τσεχία και σε σχέση με τη Unilever. Λάβατε ένα φύλλο σαν και αυτό που σας δείχνω. Προφορική τροπολογία. Unilever, εντάξει. Το βρήκατε. J'avais des idées. Eh bien oui, mais donc le femme, il faut toujours le mettre en ligne. Est-ce que tout le monde est prêt à voter Μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε. Πολύ ωραία. Ως προς την πρόταση επιστολής που εξετάστηκε από την ομάδα εργασίας. Υποβλήθηκε μία προφορική τροπολογία που υποστηρίζεται από τον κύριο Χάγκελς εκ μέρους του ΕΛΚ, την κυρία Χάρκιν εκ μέρους των Φιλελευθέρων οι πράσινοι συμφωνούν, είμαι σίγουρη, και εγώ ίδια το υποστηρίζω εκ μέρους των σοσιαλιστών. Και η κυρία Φιγκερέντο είναι πολύ ευτυχής με αυτή την προφορική τροπολογία. Σας προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το σύνολο της επιστολής όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Του Ψηφίσατε, έληξε ψηφοφορία. 46 ομόφωνα. Σας ευχαριστώ. Ψηφίζουμε τώρα. Ο κύριος Μπενάμιας. Σας υπενθυμίζω απλώς ότι η ομάδα μας είναι δημοκράτες και φιλελεύθεροι. Το όνομα δηλαδή θα ήθελα να σας υπενθυμίσω. Ναι βεβαίως όπως όλες οι ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, είναι όλες, όλοι δημοκράτες. Παντού υπάρχει το δημοκράτες. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο 29, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την Πολωνία. Υπέρ. Κατά αποχές ή διαψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Αποστέλνουμε αυτές τις δύο επιστολές στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Τώρα ερχόμαστε στην αρχική σειρά ψηφοφορίας, δηλαδή πάμε πίσω στο 18. Το 18 λοιπόν αφορά την ψηφοφορία après Έλεγα λοιπόν ότι το 18 αφορά την ψηφοφορία για την, το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Νέτζα Χίρς σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση ώστε να υποστηριχθεί η Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ευρώπη 2020. 19 τροπολογία της κυρίας Παπαδοπούλου. Υπέρ, κύριος Χάντεν. Δεν συγχωρείτε που σας διακόπτω πριν από τη ψηφοφορία, αλλά όσον αφορά τον κατάλογο ψηφοφορίας λέγεται εσφαλμένα ότι οι συμβιβασμοί γίνονται δεκτοί από την ΚΟΕ. Εμείς αντίθετα ανακοινώσαμε ότι όσον αφορά τους συμβασμούς δεν συμφωνούμε με κανέναν. Δεν υποστηρίζουμε κανέναν. Ευχαριστώ λοιπόν για τη συμβολή της ΚΟΕ για το σύνολο των συμβιβαστικών ε, τροπολογιών. Α, με την εξαίρεση όμως ε, του συμβιβασμού ε. Α λοιπόν συμβιβασμός. Περ κατά εγκρίνεται. Σημείο 26. Πολιτιστική Επιτροπή. Όπως και το 9. Γκρίθηκε. Τρία των γυναικών υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 της κυρίας Κρετή υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 23 Θέλετε να επαληθεύσουμε το 22 της κυρίας Κρετού. Ε, θα έχετε σίγουρα δίκιο. Επαληθεύουμε λοιπόν. Ψήφισατε όλοι. Έληξη ψηφοδορία 24 υπέρ, 21 κατά. Τώρα ερχόμαστε στο 23 της κυρίας Κρετού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 3.24. Τροπολογία κατάργησης υπέρ του 24, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Β. Συμβιβαστικό υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 της κυρίας Παπαδοπούλου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 του κυρίου Άλμερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τούργεν 33 εγκρίνεται Παράγραφος 5 συμβαστικό C υπέρ κατά εγκρίνεται Παράγραφος 5 Τώρα περνάμε στο 9 τη ΣΥΜΚΟ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 της ίδιας Επιτροπής. Υπέρ, κατά, αποχές, 36 της κυρίας Κρετού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 καταπίπτει. 39 υποβάλλεται ακόμη τροπολογίες. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 με προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 της ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 644 Έλμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός D. Α, θα επαληθεύσουμε το 44 κάποιος το ζητά. Ψηφίσαμε, ευχαριστώ. 21 υπέρ, 21 κατά, απορρίπτεται επόση. Συμβασμός D. Καλά κάνατε που ζητήσατε παλήθευση. D λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά το 6, 1 των γυναικών. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το 2 της ίδιας επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18. Επιτρο πολιτιστική. 15 των γυναικών μάλλον υπέρ κατά αποχές. 48 της κυρίας του Εμπεγγένη για την παράγραφο 7 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 49. Παράγραφος 7. 11 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8 το 52 υπέρ κατά αποχές δεν είναι προφανές το αποτέλεσμα και είναι και παράξενο θα έλεγα. Ψηφίσατε όλοι, έληξη ψηφοφορία. 25 υπέρ, 18 κατά, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Το 50 καταπίπτει, 51, 54 μάλλον της κυρίας Τούρμπιγεν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 του κυρίου Ποπάκη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 56 της κυρίας Τούρμπιγεν με προφορική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 57 της κυρίας Πλόντ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 των γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 της κυρίας Χίρς υπέρ κατά εγκρίνεται. 59 του κυρίου Πουπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 της κυρίας Τούρμπιγκεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 μπορούμε να το ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 των γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60, 64 ποπάκης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Συμβιβασμός ε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 11 το 9 των γυναικών. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 Πουπάκης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Εφ. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στο 8 της, των γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 Ποπάκης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 του κύριου Ποπάκη πάντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1376 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την παράγραφο 1378 του κυρίου Έλμερ με προφορική υπέρ ε, κατά απορρίπτεται. Θα το υπαλληθέψουμε εντάξει, το 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσαν όλοι, έληξε ψηφοφορία. 21 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, Κάτι λέγεται από κάτω χωρίς μικρόφωνο. Από την ώρα που θα ψηφιστεί από την Επιτροπή θα είναι η θέση της Επιτροπής. Συνεπώς το όνομα δεν θα αναφέρεται. 79 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 των γυναικών υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην παραγράφο 14G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 της κυρία Παπαδοπούλου υπέρ κατά εγκρίνεται 83 του κυρίου Ούγκορλενού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 Πουπάκης υπέρ κατά απο, εγκρίνεται 85 υπέρ κατά εγκρίνεται 86 υπέρ κατά εγκρίνεται 87 υπέρ κατά εγκρίνεται. 88 ε, Handel υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 Τούρμπιγκεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 τη ΣΥΜΚΟ με προφορική τροπολογία των πρασίνων δεν υπάρχει αντίθεση. Ε, όπως τροποποιείται ψηφίζουμε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 πλόμ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 17. H. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18. 96. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 χιρς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 Πουπάκης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 ή υπέρ κατά εγκρίνεται και τώρα ερχόμαστε στο 8 της ΣΥΜΚΟ το 2 της ίδιας επιτροπής εγκρίνεται Παράγραφος 20G. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Τη ΣΥΜΚΟ πάντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά από την 20, την 106 του κύριου Φουπάκη, προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21, 107, 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 κυρία Παπαδοπούλου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 του κυρίου Ποπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παραγραφός 23, η 10 Επιτροπής Γυναικός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 ε, ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 και 23 εντάξει θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί 112 της κ. Παπαδοπούλου υπέρ 111 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 Έλμερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 Επιτροπής Γυναικών υπέρ 113 του κ. Έλμερ, 113. Και αν ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. 22-24. Δίκιο έχετε. Απορρίπτεται. 5 επιτροπές γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 της Ροντζόλη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 επιτροπές γυναικών υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται, 115 κύριε Τουρίν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 1 Τουρίν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, α το κάπα το υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, α Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, β Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 Τούρινεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 Έλμερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το Β Ελ. λατινικό συμβαστική λύση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το Σ, το ΕΜ. το λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 Έλμερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 του κ. Ποπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για να δούμε τώρα τελική ψηφοφορία το ψήφισμα αυτό. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Και ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 43 υπέρ, ένας κατά και τρεις αποχές. Συγητή για τον εισηγητή μας συγχαρτήρια. Πάμε παρακάτω. Γιούτα Στάρκ, Επιτροπή για το θέμα της 1α ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1, τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 1, τρο... Β υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται από 1. Το γάμα το λατινικό, το, συγγνώμη, το λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. παραφώς 2. Ε, ε το λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία F, λατινικό, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3, το G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3, τροπολογία 43, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 4, τροπολογία συμβαστική H, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παραγραφός 4, τροπολογία 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παραγραφός 4, τροπολογία συμβαστική Ή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 68, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69, υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Παράγραφος 5 τροπολογία συμβαστική Ζ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5 δύο τροπολογίες ταυτόσιμες 90-91 ψηφίζουμε και τις δύο μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 5 τροπολογία 6, η 96, λιν, υπέρ, κατά, αποχές, κανονικά εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Και αν ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας, για να δούμε. Γρήγορα, γρήγορα. Πέρας ψηφοφορίας λοιπόν, 32 υπέρ, 14 κατά, Πλατεία πλειοψηφία ψήφισε υπέρ, η 4 καταπίπτει. Την 6, 107 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ, κατά. Δεν ψηφίσατε. 108 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 110 του κύριου Πουπάκη Μια παρατήρηση εκτός μικροφώνου, ότι κάποιος, αν ακούμε καλά, δεν μπόρεσε να ψηφίσει, δεν ψήφισε. 96. Κάλυπτε όμως ε, το σύνολο της βασική λύσης κάπα λατινικό. Δίκιο, δίκαιο, δίκιο, δίκαιο έχετε και με συγχωρείτε. Απόλυτα δίκαιο. 106 King ναι, που συνδυάζεται με την 96 λίν. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 του κύριου Πουπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 το L το λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τα την 7 έχουμε την τροπολογία 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μισό λεπτό, μισό λεπτό κάτι. Το ίδιο αντιμετωπίζουμε και εδώ όπως πριν. Με την 121 μπακ. Μετά την παραγραφό 7. 121 μπακ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και συγγνώμη. 122 όχι. Λοιπόν και 123 του κύριου Μπουπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8. Συμβαστική εμ λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά από την 8, 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τον 37 να ψηφίσουμε στη συνέχεια. Θα δούμε τι γίνεται τώρα. Το πει το λατινικό θα ψηφιστεί, θα υπερψηφιστεί όχι. 9, εν λατινικό υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Πού πάμε τώρα, μετά την 9, παράγραφο, τροπολογία ο συμβαστική. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μετά την νέα 152 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 153 του κ. Ποπάκη ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10 τη συμβαστική π υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 137. Μετά την 10 έχουμε την 163 Ροντζόλη υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται παράγραφο 11 συμβαστική ε, Q υπέρ. Κατά αποχέ ε, εγκρίνεται. Και μετά την 11 παράγραφο 172 Γιώτοβα με προφορική τροπολογία. Δεν είναι κανείς αντίθετος αυτό. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 11 έχουμε την 173 στα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11 το R συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την 11 έχουμε την 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 178 2 υπέρ κατά αποχές το ίδιο απορρίπτεται 179 του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ κατά αποχές 181 καταπίπτει αυτή ψηφίζουμε λοιπόν 182 και 193 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 184 υπέρ κατά αποχές κανονικά απορρίπτεται. Να δούμε, να δούμε ηλεκτρονικά παρακαλούμε. E Και πάλι πολύ πολύ από το ΕΛΚ. Ah, alors, euh, Πέρας ψηφοφορίας κανονικά, ναι. 28-18 το αποτέσμα. Εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 186 υπέρ. Κατά αποχές γκρίνεται. Ψηφίζουμε ε, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονική ψηφοφορία, το σύνολο του κειμένου. Τώρα δεν έχει πολλού από το ΕΛΚ. Όχι κύριε Μπορέν, δεν, δεν έχετε δικαίωμα να ψηφίσετε. Τι να σας πω, δικό σας το πρόβλημα, στον οίκο σας. Λοιπόν, τι έγινε, ψηφίσαμε. πέρα ψηφοφορία. Ήρεμα, ήρεμα, μπορούμε να ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορία. Έτσι κι αλλιώ σχεδόν όλοι ψήφισαν υπέρ. Μην ξαναρχίσουμε να ψηφίζουμε τώρα. Υπέρ 41, κατά 4, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια μας. Πάμε παρακάτω. Σημείο 20. Ένωση καινοτομία μεταμορφώντα την Ευρώπη για ένα κόσμο μετά την κρίση. Σαρή Εσαγιά. Η συντάκτρια. Alors, paragraphe 1. 1α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παραφάσα 1 τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 τρο... της υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να την 1 τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παραφάσα 2 το β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3, την γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3, τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. εγκρίνεται. Παραφός 3, τροπολογία 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Να, ψηφ... να ελέγξουμε την 20 αν θέλετε. Ψηφίστε το όλοι, έλξη ψηφοφορία. Έλξη. Ωραία. 21 υπέρ, 23 κατά. Έχετε δίκιο. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 σε δύο μέρη. Το σύνολο της τροπολογίας εκτός το ΒΕΡ θα ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ χωρίς το ΒΕΡ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ποιος θέλει τώρα να προσθέσει και το ΒΕΡ. Ποιος δεν θέλει να το προσθέσει. Ποιος απέχει. Λοιπόν, προσθέτουμε και τους πρασίνους. Α, επαλήθευση, ωραία. Λοιπόν, εγώ ψηφίζω υπέρ των πρασίνων. Ψηφίζατε όλοι. 21 πουρ. 21 υπέρ, με συγχωρείτε, 24 κατά. Δεν λειτουργήσε. Κύριε Έλμερ. Δεν θέλω να επικρίνω, αλλά λέτε ποιοι είναι υπέρ, μετά κοιτάτε χαμηλά τα μάτια σας και μετά λέτε ποιοι είναι κατά. Και δεν μπορούμε να προλάβουμε για, να, για τη διεξαγωγή της, τη σωστή αυτής της ψηφοφορίας. Ε, είχαμε δύο τέτοια παραδείγματα, το ένα μετά το άλλο, όπου είπατε ότι υπερψηφίστηκε ε, ενώ τελικά βγήκε ότι καταψηφίστηκε η τροπολογία. Παρακαλώ, θα ήταν πιο ευγενικό από εσά εάν κοιτάτε τα μέλη όταν ψηφίζουν υπέρ κατά και όχι να χαμηλώνετε τα μάτια. Βεβαίως δεσμεύομαι κύριε Έλμερ και να κοιτάω και να υπαλληθεύω. Ε, λοιπόν, επανερχόμαστε. Συμβιβαστικό δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, τροπολογία 26 σε δύο μέρη, η κυρία Εσέρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει ένα λάθος στον κατάλογο ψηφοφοριών, δηλαδή έχει γίνει ο διαχωρισμός με λάθος τρόπο. Θα πρέπει να κάνουμε το εξής. μέχρι τις λέξεις που αφορούν το περιβάλλον, μέχρι εκεί να είναι το πρώτο μέρος της ψηφοφορίας και εν συνεχεία το δεύτερο. Στον κατάλογο ψηφοφοριών του ΕΛΚ θα πρέπει να υπάρχει συν και όχι μείον. Αντί λοιπόν να μιλάμε για λέξεις, χωρίζουμε την τροπολογία σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος και δεύτερο μέρος. Το ΕΛΚ είναι υπέρ του πρώτου μέρους και του κατά του δεύτερου μέρους. Δεν μπορώ βεβαίω να ανακοινώσω την τοποθέτηση των άλλων ομάδων, δεν τη γνωρίζω, αλλά δεν σας καλώ βέβαια να το δηλώσετε δημόσια. Πρώτο μέρος λοιπόν, μέχρι την λέξη 2002. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ του υπόλοιπου κειμένου. Υπέρ, κατά, αποχές θα το επαληθεύσουμε. Tout Όλοι υπέρ, κατά, δεν εγκρίνεται το δεύτερο μέρος. Τροπολογία 27, γκοντζούλη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 του κυρίου Πουπάκη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 του ίδιου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 Ισαΐα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 της κυρίας Σέτερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κρίνεται. Ο κύριος Έλμερ ήταν κατά. Τροπολογία 35 Κρουντζόλη με προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Σρέτερ. Παράγραφος 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα υπαλληθεύσουμε. 37 Σρέτερ. 36 ε, λέει τώρα η πρόεδρος. Αρχιετή ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται το σαφήνεια. 38 μεσάγια υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 μεσάγια υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40. Κροντζούλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 41 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 42 κροντζούλη υπέρ κατά εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα του κειμένου ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσαμε, έληξη ψηφοφορία. 45 υπέρ, 0 αποχές, 0 κατά ομόφωνα. Συγχαρητήρια κυρία Συγγήτρια. Και τώρα περνάμε στο 21. Πρόκειται για την έκθεση για την ενίσχυση της εποπτείας της μεσονομικής κατάστασης. Έχουμε δύο τροπολογίες που από την κυρία Φιγκυρέντο, το Ράντελ Τσίμερ και για Ρίκ. Τα ψηφίζουμε μαζί. Πρόκειται για τις τροπολογίες 64, 63, 64 υπέρ κατά απορρίπτονται. Σύνολο του κειμένου. Προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για το σύνολο του κειμένου έχουμε και συμβιβιστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 1 Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 με προφορική της εισηγητρές. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 της γήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 της γήτριας υπέρ κατά α, θα επαληθεύσουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έλξη ψηφοφορία. 23 υπέρ, 20 κοτά, εγκρίνεται. Άρθρο 1. Σημείο 2. Συμβιβαστικό F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστικό G. Ποιος υπέρ κατά 21 εισηγητού υπέρ κατά 22 επίσης του εισηγητού υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστικό H. Υπέρ. Υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Συμβαστική H λοιπόν. Ψήφισαν όλοι. Έληξη ψηφοφορία. 21 υπέρ, 21 κατά, 4 αποχές. Δεν εγκρίνεται. 24 της υπέρ. Με συγχωρείτε, λάθος. 24 έχει περάσει. Καλύπτεται μάλλον. Απορρίψαμε με τον συμβιβασμό. Πάμε στο 88. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε το 23. Ψηφίσαν όλοι. Ευχαριστώ. 40 υπέρ, 6 κατά. Εγκρίνεται. Το 89 καταπίπτει. 24 έχει καταπέσει. Και, και, και, και. Το 90 επίσης. Και έτσι ερχόμαστε στην τροπολογία 25 της ηγετρίας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να το 25. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε. Έληξη ψηφοφορία. 22 υπέρ, 22 κατά, μία αποχή δεν εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία. Όχι. Τροπολογία 91 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία τη συμβιβαστική ή, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας επαληθεύσουμε το 27. Ψήφισα τα όλοι. Έληξη ψηφοφορία. 21 υπέρ, 23 κατά, απορρίπτεται. Η τροπολογία 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε το 90, την 95. Έλξη ψηφοφορία. 37 υπέρ 5 κατά. Εγκρίνεται, σαφέστατα. Άρθρο 1 σημείο 4J. Υπέρ. Ναι, κύριε Χάντελ. Κύριε Πρόεδρε, ε, υπό το J, ο Τόμας Χάντελ και η Γκάμπριελ Τσίμερ την, τον, έχουν τα ονόματά τους. Εμάς δεν μας ρώτησαν ε, εάν θέλουμε να διαγραφούν τα ονόματα ή όχι. Um, Euh, Κύριε Χέντελ, μου κάνει εντύπωση το ότι δεν ζητήθηκε η άποψή σας. Εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνομαι την απόσυρσή σας από τη συμβαστική συνεπώς ο, ο κύριος Κάζα εκ μέρους της, του ΕΛΚ το υποστηρίζει. Ε, ψηφίζουμε τη συμβαστική λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ερχόμαστε στην τροπολογία 97 του κυρίου Καζάκ υπέρ κατά κατά αποχές θα επαληθεύσουμε δεν είδα καλά το κατά ψηφίσατε όλοι έληξη ψηφοφορία 22 υπέρ 24 κατά δεν εγκρίνεται κα συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλα συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ερχόμαστε στη συμβιβαστική έμμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο όμικρον συμβαστική πάντα υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε τη συμβαστική όμικρον και αν ψηφίσατε πέρα ψηφοφορία 22-23 για μία ψήφο απορρίπτεται τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 γιγκολιπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 36 καλύπτεται 108 και αυτό και αυτή Επόμενη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 ορί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 ψηφίζουμε υπέρ της 38 να ελέγξουμε αν θέλετε για την 109 υπέρ ε, κατά κατά λοιπά, Και αν ψήφισαν όλοι. Για την 109, 109 ψηφίζουμε κύριε Αλμέρ. Τροπολογία 109. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 19-26. Απορρίπτεται. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 111 με προφορική τροπολογία Κρόιτσμαν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 40 εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 41 εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. 41, 41. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 22-21 εγκρίνεται. Δύο οι αποχές. τι είπατε εσείς. Ναι, 22-21. Δύο αποχές εγκρίνεται. Το π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 45. 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. R λατινικό υπέρ. Απορρίπτεται η 45. Να ελέγξουμε. Η R, όχι η R, R. Λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά πίπτη 45. Πού πάμε τώρα. 48. Υπέρ της 48. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε για τη 48. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας, 22-23 απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 116 Γκίγκολτ υπέρ. 116 κατά αποχές εγκρίνεται. 49 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 του ιδίου υπέρ. Κατά αποχές. Κανονικά απορρίπτεται να ελέγξουμε όμως. Και αν ψήφισαν όλοι, ψηφοφορια ψηφοφορίας. 41-5 εγκρίνεται. 52 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 118 καζα υπέρ. Κατά. δεν βλέπω καθαρά ποιο είναι το αποτέλεσμα. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία και αν ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 22-24 απορρίπτεται. Το επόμενο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 54 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το ταφ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το U υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εξήντα τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε την 58. Ποιοι είναι υπέρ της 58. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα η τροπολογία 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ναι, 127 να ελέγξουμε αν θέλετε. 127 ελέγχουμε. 127 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Και αν ψήφισαν όλοι πέρα τις ψηφοφορίες, 19, 27 κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 2 του εισηγητή. Όχι, όχι. Την ένα, την ένα. Την ένα του εισηγητή ψηφίζουμε. Την ένα, υπέρ. Μισό λεπτό, μισό λεπτό ε, βλακίες κάνω. 61, 61. Ψηφίζουμε για την 61. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα τώρα. Ένα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ αποχές εγκρίνεται 65 γίγκολτ με προφορική τροπολογία 66, 66, 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4 του εισηγητού και πάλι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά από την 5, τη β, τη συμβαστική υπέρ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τη γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. οκτώ τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η εννέα τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 γίγκολτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τη δέλτα βαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ 12 την ε τη συμβαστική υπέρ κατά την ε υπέρ είπαμε κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλούμε υπέρ και υπέρ κατά λοιπά Ναι, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Και αν ψήφισαν όλοι, Πέρας ψηφορίας. 35 υπέρ, 2 κατά, οι αποχές 6. Το δεύτερο κείμενο, χειροκροτήματα, ευχαριστώ. Έκθεση Κάζα. υπερβολικά ελλείμματα, τρει ταυτόσιτε με 21-22 κλπ. 20-21-22 υπέρ κατά απορρίπτεται. απορρίπτεται. κυρία Ήρς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι εμείς ως φιλελεύθεροι υποστηρίζουμε οπωσδήποτε τη συμβιβαστική Α. Σας ευχαριστούμε για τη διευκρίνησή σας. Να σας πω κάτι. Για τις συμβεστικές τροπολογίες είμαι γεγραμμένος. Ε, δεν είμαι, δεν είμαι σε αυτές. Ε, τεχνικό το λάθος. Εντάξει, εντάξει. Το σημειώνουμε. Καταπίπτει η α συμβαστική, πάντως οι φιλελεύθεροι το υποστηρίζουν, άρα λοιπόν μπορεί έτσι κι να ψηφιστεί, αλλά σας ευχαριστούμε για τη διευκρίνησή σας φιλελεύθερη και δημοκρατική ονομάζεται η ομάδα μας. Να το υπενθυμίσω. Εντάξει, αν θέλετε να σας πω και μια ιστοριούλα θα σας το πω όμως μετά την ψηφοφορία. Για το σύνολο τώρα του κειμένου, τι έχουμε. Έχουμε μια τροπολογία προφορική που ψηφίζουμε. Οριζόντια, οριζόντια. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 γκίγκολτ σε δύο μέρη χωριστά. Θα σας ταράξει αν το κάνω ανάποδα. Γιατί κανονικά πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα χωρίς αυτές τις λέξεις, έτσι αυτό ότι θα έπρεπε να μειώνεται κάθε τρεις, ε, τρία χρόνια. Ε, χωρίς αυτή τη φράση ψηφίζουμε υπέρ. Ε, μάλλον κατά. Αποχές. Απορρίπτεται άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτό ή μήπως όχι. Κύριε Γκίγκολ, τι γίνεται. Χρειάζεται να ψηφίσουμε, ε, έχει νόημα το υπόλοιπο του κειμένου. Εντάξει, συμφωνείτε, τι κάνετε. Όχι, ψηφίζουμε και το υπόλοιπο, υπέρ. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι μισό λεπτό μέχρι το ποσοστό χρέους που θα πρέπει να μειώνεται κάθε τρία χρόνια κλπ. Περκατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 κάζα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 μπορεί να συνδυαστεί υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Όχι. Α, απορρίπτεται, απορρίπτεται, απορρίπτεται. 32 Γίγκολτ ε, σε δύο χωριστά μέρη. Πρώτο μέρος. Η Επιτροπή μέχρι το Συμβούλιο. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου μέρους της τροπολογίας του κ. Γίγκολτ, Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος τώρα, το επόμενο κείμενο, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μπορεί να συνδυαστεί 33, την ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 τροπολογία για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 35 γκίγκολτ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία συμβαστική από τους φιλελεύθερους και δημοκράτες. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται η Β, η συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 11 του κυρίου Κάζα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τη 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 γκλουτς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 όχι συγγνώμη 44 44 44 κανονικά ναι, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 του εισηγητή 14 λέγω ψηφίζουμε υπέρ υπέρ της 14 κατά αποχές εγκρίνεται 45 γλούτς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 του ιδίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 18 του εισηγητή με τεχνική διόρθωση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 καταπίπτει πάμε στο, στην στη συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά δεν είναι σαφές. Υπέρ για τροπολογία 1. Τώρα είναι σαφές. Ευχαριστώ. 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. γίγκολτ, Το 26 υπέρ κατά εγκρίνεται. 3 καζάκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 καζάκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 ε, εγκρίνεται 23 στο 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 24 υπέρ κατά απορρίπτεται 25 γκίγκολτ υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω. Θα το απαλληθεύσουμε. Ίσως να απορρίπτεται, αλλά δεν είναι και σίγουρο. Ψηφίσατε. Έλεξη ψηφοφορία. 18 υπέρ, 23 κατά, απορρίπτεται. Σκέψη 12, τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου τώρα, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έληξη ψηφοφορία 39 υπέρ, 4 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Τώρα περνάμε στη δεύτερη έκθεση Καζά που έχει να κάνει με την ενίσχυση της εποπτείας της μουσιονομικής κατάστασης. Ε, τρεις τροπολογίες κατάργησης, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Ε, τροπολογία 10 του εισηγητή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 30, με προφορική, υπέρ, κατά, αποχές, επαληθεύουμε το, την 30. Ψηφίσατε όλοι. Έλξη ψηφοφορία. 36 υπέρ. Εγκρίνεται σαφέστατα. 32. Με προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 του εισηγητή. Με προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 37 μπλουτ με δύο μέρη. Εδώ θα αντιστρέψουμε την ψηφοφορία. Το κείμενο χωρίς and after consulting the parliament. Το σύνολο λοιπόν του κειμένου εκτός αυτών των λέξεων. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 Κρόιτσμαν υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Επαληθεύουμε την 36. Ψηφίσατε 23 υπέρ, 20 κατά. ε, γκρίνατε, με συγχωρείτε. 12 του εισηγητή Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40. Πλούτς. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42. Γλούτς, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 Κρότσμαντ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 του εισηγητή με προφορική. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 Γκλουτς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 7 συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στην τροπολογία 1 του εισήγητη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σκεπτικό 3 συμβαστική α υπέρ κατά εγκρίνεται. Τρεις τροπολογίες για το β υπέρ κατά εγκρίνεται. 21 γκίγκολ με προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 5 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 γκλουτ με προφορική υπέρ κατά αποχές. Η τροπολογία 23 καταπίπτει, με συγχωρείτε και η 6. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε την 6. Τροπολογία 24 την ψηφίσουμε γιατί η 36 κρίθηκε. 24 δηλαδή. Υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Σκεπτικό 5, τροπολογία 25 με προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 9, τροπολογία 29, Κρότσμαν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 11, συμβιβαστική C, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 τροπολογία 9 του συντάκτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου τώρα ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έληξη ψηφοφορία. 36 υπέρ, 4 κατά, 4 αποχές. Συγχαρητήρια και πάλι στον εισηγητή. Ερχόμαστε στη τρίτη έκθεση του κυρίου Καζά. Τρεις προτάσεις απόρριψης πρόσκειται για την έκθεση για τη το δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Άρθρο 1. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6. Του συντάκτη. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16. Με προφορική. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 του συντάκτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 του συντάκτη πάντα υπέρ έκανα λάθος ψηφίσατε το ένα, το αμφισβητήσατε πρέπει να πάω πιο σιγά. Δύο λοιπόν, δύο. Τροπολογία δύο. Κατά. Ε, εγκρίνεται. Τρία. Ε, ε, μπορεί να συνδυαστεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έντεκα τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου ψηφίσατε όλοι. Έληξη ψηφοφορία. 41 υπέρ. 4 κατά και μία εποχή. Ο κύριος Καζά έχει όλο και καλύτερη βαθμολογία στον συγχαρούμενο λοιπόν. Και τώρα φτάνουμε στην πρώτη τελευταία μας ψηφοφορία για την πρόληψη και την διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Τρεις τροπολογίες κατάργησης. 43, 44, 45. Υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Άρθρο 1, τροπολογία 24. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 2, ε, συμβαστική H. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πολύ γρήγορα πήγα, συγγνώμη. Το H λοιπόν, συμβιβαστική H. Ψηφίσατε. Έληξη ψηφοφορία. 22 υπέρ, 23 κατά. Έχετε δίκιο, απορρίφθηκε. 57-59 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 25 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 2058 με προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβιβαστική ή υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έλξη ψηφοφορία. 22 υπέρ, 24 κατά. Δεν εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 26 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. G συμβιβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται. K υπέρ κατά εγκρίνεται. 67 του κύριου Γκίγκλς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλα συμβιβαστική διακοπή. Ψηφίσατε όλοι. Έληξη ψηφοφορία. 22 υπέρ, 23 κατά, απορρίπτεται με μικρή ψηφοφορία. Συμβαστική έλα υπέρ, κατά. Εγκρίνεται, σας το υπόσχομαι. 30 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έμμα συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ κατά εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές Α, νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά να το απελευθεύσουμε. 81 ψηφίζουμε. Έληξη ψηφοφορία 22 22 υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά. Αποχές Κανείς δεν ψηφίζει πια. 34. Ξανά. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82. Γκλουτσκι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35. Εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83. Με προφορική. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 του εισηγητή. Υπέρ 83 ζητάτε επαλήθευση. Αν αλλάζει η γνώμη το ΕΛΚ, ε, τέλος να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσαμε. 27-19 εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το πι, συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε το πι ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 19-24, δύο οι αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 84 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 37 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 85 σε δύο μέρη χωριστά χωρίς το σαλ αυτό το θα ποιος είναι υπέρ του κειμένου χωρίς το θα έπρεπε ε, υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται δεν χρειάζεται να ψηφίσουν το υπόλοιπο λοιπόν 38, 36, 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 γλουτς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40, 92, 96 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 41, 93, 97 ταυτόσημες ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 42, 94, 98 ταυτόσημες ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 99, 95 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Να δούμε, να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. 95-99. πέραση ψηφοφορίας. 27-18 εγκρίνονται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 2 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται α στην τελική σκέψη 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά από το 6 την συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την τα τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 ναι, συνδυάζεται υπέρ κατά αποχές ε, κανονικά απορρίπτεται να το ελέγξουμε όμως. Παράξενο μου φαίνεται να απορρίπτεται αλλά να το δούμε, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας 29 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι δύο οι συμβαστικοί υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η εφ συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 20 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η G, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου τώρα, η ηλεκτρονική ψηφοφορία βέβαια. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρα της ψηφοφορία. 36 υπέρ, 2 κατά, οι αποχές 8. Και τώρα τελευταία ψηφοφορία. Προτελευταία, προτελευταία ψηφοφορία. Ουχή τελευταία. Non, non, non. Non, j'invite <laughs> Εντάξει, να αλλάξει κανεί όσον αφορά τη ψηφοφορία. Να αλλάξουν και διάθεση. Ψηφίζουμε την τελευταία έκθεση για τη διαχείριση, διακυβέρνηση. Μακροοικονομική πειθαρχία. 18-19 διαγραφής ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 13 ψυχή υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 30 τροπολογία έτοιμο για ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρος. Το bargaining structure. Αυτό. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου μέρους. υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν έχει νόημα τώρα να ψηφίσουμε το δεύτερο μέρος αφού απορρίφθηκε το πρώτο. Να ψηφίσουμε αν θέλετε το δεύτερο μέρος της 30 τροπολογίας. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 και 32 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά δεν βλέπω να είναι σαφές το αποτέλεσμα. Να ψηφίσουμε για το 16 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Ναι, ναι, ναι, τα μπέρδεψα να ξαναρχίσουμε. Τροπολογία 16. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά πάλι την 16, για τη 16. Ψηφίσατε πέρας ψηφοφορίας. Να ψηφίσουμε. Κάποιος, κάποιοι ψήφισαν παραπάνω. Να ψηφίσουμε για τρίτη φορά. 16. Ψηφίζουμε ξανά τρίτη φορά για την 16. Ένας από το ΕΛΚ ε, είναι παραπάνω. Ψηφίσατε. Ναι, πέρασε φορείας και 16-22-22 απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 μπορεί να συνδυαστεί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η Β συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κάποιο λάθος υπάρχει. Το 146 αντιστοιχεί με το 148 κανονικά. Ε, τι να σου πω. Το διορθώσουμε μάλλον. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 26-27 ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 τη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου τώρα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 37 υπέρ, κατά 4, οι αποχές 6. Τελειώσαμε λοιπόν με την ε, οικονομική διαχείριση. Ε, τον συνεισηγητή μου, τον κύριο Κάζα, τον ε, συγχαίρω, τον ευχαριστώ. Διεργαστήκαμε και τώρα τελευταία ψηφοφορία. Αλεσάνδρο Σέρκας. Διαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας. 1β, 14 τροπολογία. Ομεν Ρόιτεν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 τροπολογία για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 Λαμπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25-26 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 27-28 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 34-35 ταυτόσημες ψηφίζουμε υπέρ. Μάλλον είναι διαγραφής αυτές. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 36-37 για διαγραφή ταυτόσημες ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Άρθρο 12, παράγραφος 2, δέλτα, 38 τροπολογία σέρκα. 39 Λογιάρικ, 40 ΟΜΕΡΟΙΤΕΝ, Ρόιτεν. για διαγραφή, ψηφίζουμε υπέρ τη διαγραφή κατά απόχέ εγκρίνονται. 41 αποσύρθηκε, αλλά έτσι κι αλλιώς καταπίπτει, έτσι. 42-43 ταυτόσιμες, ψηφίζουμε 42-43, για διαγραφή είναι, υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Και ψηφίζουμε τη δέλτα τη συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Τη δέλτα 1. Τη δέλτα 2 τώρα συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 Omen Reuten. με προφορική τροπολογία με το από πλευρά κρατών μελών ε, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές. Να λέξουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία 52 του εισηγητή. Nous votons l'amendement 52 de... 52 του κυρίου Σέρκας. 52 του κυρίου Σέρκας. Άρθρο 13 παράγραφος 2. Καινούριο εδάφιο. Ψήφισα το όλοι εντάξει. Ευχαριστώ. «21 υπέρ, 25 κατά, μία αποχή δεν εγκρίνεται». Τροπολογία 1. Μεσάια υπέρ κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το επαληθεύσουμε. Ψηφίσατε, έληξη ψηφοφορία. «26 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται». Το 2 καταπίπτει. Το 3. Ο Ιμεν Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Ομένο Υπέρ, α, τέσσερα με συγχωρείτε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 της ίδιας. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7. Ίδια συντάκτρια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 μεσάια. υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο πληθεύσουμε καλύτερα. Ψηφίσατε όλοι. Έλξη ψηφοφορία. 26 πέρ 21 κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα μετά το 16 στην τροπολογία 9 της Όιμεν Ρόιτον με προφορική για την κατάργηση του μίνιμουμ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 σέρκας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ερχόμαστε ηλεκτρονικά στην τελευταία ψηφοφορία ψηφίζουμε ψηφίσατε όλοι έληξη ψηφοφορία ε, πολλοί πάλι ψηφίζουνε Ξαναρχίζουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Ξαναρχίζουμε επαναλαμβάνω. Δεν ήταν η τελευταία μας αυτή. Κυρία Όιμεν Ρόιτερ, ψηφίζουμε. Είναι η τελική ψηφοφορία. Υπήρξε ένα σφάλμα. Ψηφίσατε όλοι. Έλξη ψηφοφορία. 33 υπέρ, 12 κατά, μία αποχή. Συγχαίρουμε τον εισηγητή μας. Θα ήθελα να ζητήσω από όσου φεύγουν από την αίθουσα να το πράξουν ήρεμα και χωρί συζήτηση. Κύριε Κάστλερ, κύριε Κάστλερ, σας παρακαλώ να μην φύγετε από την αίθουσα, διότι έχουμε εγκρίνει την έκθεσή σας και ενδεχομένως πρέπει να υπάρξει μία διαπραγμάτευση κατά την πρώτη ανάγνωση για να υπάρξει συμφωνία. Λοιπόν, υπάρχει πολύ φασαρία στην αίθουσα δυστυχώ, διακόπτει πρόεδρος. Bien. Monsieur um, Κύριε Κάσλερ κανονικός εγώτων των πραγμάτων. Πρέπει να ξεκινήσουμε μία διαπραγμάτευση για μία πρώτη ανάγνωση. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχετε εντολή από την Επιτροπή. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή το εξή. Λίγο σεβασμό σας παρακαλώ. Πρόκειται για νομοθετικό έργο. Θα δώσουμε εντολή διαπραγμάτευση στον κύριο Κάσλερ και σε μένα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Ζητώ τη γνώμη σας, παρακαλώ. Συμφωνείτε να μας δώσετε αυτή την εντολή, αυτή την εξουσιοδότηση, ώστε να αναζητήσουμε συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση, με βάση την ψηφοφορία ε, που είχαμε σήμερα το πρωί. Μοιάζεται να συμφωνείτε, σας ευχαριστώ και θα ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης. Και τώρα ερχόμαστε στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι δημόσια ακρόαση για το ρόλο και τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Σητώ συγγνώμη από τους προσκεκλημένους μας για την καθυστέρηση με την οποία ξεκινάμε αυτή την ακρόαση. Αλλά νομίζω αντιληφθήκατε πόσες ψηφοφορίες είχαμε να κάνουμε σήμερα το πρωί. Πρωτού σας δώσω λοιπόν το λόγο, θα ήθελα σύντομα να ζητήσω από την εισηγήτριά μας κυρία Μωράν Σαρτιέ να μας κάνει μία εισαγωγή για αυτή την ακρόαση. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης θα ακούσουμε εκπροσώπους διαφόρων ε, κοινωνικών εταίρων. Κυρία Μωράν Σαρτιέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ ζητώ συγγνώμη από τους εταίρους μας που πρόκειται να ακούσουμε σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να σας πω πόσο σημαντική είναι αυτή η ακρόαση. Θέλουμε σήμερα το πρωί μαζί με τους κοινωνικούς μας εταίρους να συζητήσουμε το ρόλο και τις επιπτώσεις του ΕΚΤ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στον καθένα εδώ ότι το Ταμείο Συνοχής στο ευρωπαϊκό επίπεδο στο κοινωνικό τομέα αντιπροσωπεύει ένα πολύ σημαντικό τομέα. 22% των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής αφιερώνονται στην κοινωνική συνοχή ακριβώς. Η κρίση που έχει πέσει πάνω στην Ευρώπη μας αναγκάζει να, είμαστε, να ακόμη περισσότερο όσον αφορά την εξέλιξη του ΕΚΤ. Αυτή η εξέλιξη στη πορεία. Έχει σαν στόχο βεβαίως τη μείωση των κοινωνικών ανισορροπιών, αλλά καταπολεμά και την ανεργία. Και αναφέρομαι ειδικότερα στην ανεργία των νέων, που σήμερα ανέρχεται περίπου σε 23% για τις ηλικίες 18 με 25 ετών. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε και όλα τα δημογραφικά, τα πληθυσμιακά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει έως το 2020. Ε, ακόμη θέλω να αναφερθώ και στην εξέλιξη της απασχόλησης που θα πρέπει να υποκινηθεί. Σύμφωνα με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ στη Θεσσαλονίκη είναι ένας οργανισμός τον οποίο επισκεφθήκαμε με την κυρία Παπαδοπούλου και την κυρία Ήρς. Ε, λοιπόν, είδαμε ότι μέχρι το 2020 15% των θέσεων με χαμηλά προσόντα θα εξαφανιστούν, ενώ θα χρειαστούμε 5% παραπάνω θέσεις εργασίας με υψηλά προσόντα. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν μας αναγκάζει να προσδιορίσουμε σε βάθος πολιτικές για να μπορέσουν οι μισθωτοί να εξελιχθούν και να μην έχουν να αντιμετωπίσουν και νέα προβλήματα ανεργίας, ε, τουλάχιστον στις πιο εύστραστες κατηγορίες. Λοιπόν, πρέπει να οικοδομήσουμε μία συνεπή κοινωνική Ευρώπη μέσα σε ένα πλαίσιο ανταγωνιστικής αγοράς. Αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι πολύ σημαντικός μοχλός για την κοινωνική πολιτική της Ευρώπης. Και συνεπώς θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό, διότι το ΕΚΤ είναι ένα εργαλείο συνέπειας για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Είναι ένα εργαλείο κοινωνικής συνοχής, επαναλαμβάνω δεν μπορεί να απομακρυνθεί, δεν μπορεί να απεξαρτηθεί αν θέλετε από τις εθνικές πολιτικές και ξέρουμε πολύ καλά ότι η εφαρμογή του για να είναι αποτελεσματική, για να είναι τα αποτελέσματα ισχυρά πρέπει να, να έχει σοβαρή αγκύρωση και στο τοπικό και στο περιφερειακό. Έχουμε λοιπόν διάφορα θέματα που πρέπει να σκεφτούμε σε σχέση με την εξέλιξη του ΕΚΤ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν σήμερα το πρωί καλέσαμε μεγάλες ευρωπαϊκές οργανώσεις, ε, κοινωνικούς εταίρους ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Την Business Europe, την ETUC, την CEP, την UEAPME, e, τη CRPM που είναι ε, η συνδιάσκεψη των ε, θαλασσίων περιοχών, παράκτιων περιοχών και την κοινωνική πλατφόρμα, ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε από τους χρήστες πλέον πώς αντιλαμβάνονται τα προβλήματα τα οποία τίθεται στο επίπεδο του ΕΚΤ. Πώς βλέπουν δηλαδή την μελλοντική εξέλιξη ώστε να έχουμε βελτίωση των αποτελεσμάτων για μας δεν τίθεται θέμα οι ευρωπαϊκές πολιτικές να εξαπλώνονται στην Ευρώπη χωρίς να είναι αποτελεσματικές επιτόπου. Δηλαδή, για μας το σημαντικό δεν είναι να εξετάσουμε την ποιότητα της διαχείρισης αυτών των ταμείων, αλλά θέλουμε περισσότερο να μάθουμε κατά πόσο βοηθούν τον χρήστη. Γι' αυτό θα ακούσουμε τους εταίρους μας σήμερα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μαρζένα Τσιλιεύσκα της Πολωνικής Συνομοσπονδίας ε, Ιδιωτών Εργοδοτών. Σας παρακαλώ να συντομεύσετε κατά δύο λεπτά την ομιλία σας. Δηλαδή πέντε λεπτά είναι στη διάθεσή σας. Πολύ λυπάμαι για αυτή τη σύντμηση του χρόνου. Uh, Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σε αυτή την ακρόση. Συνήθως εργάζομαι σε εθνικό επίπεδο εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους και σε διάφορες εποπτικές επιτροπές για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Θα ήθελα να αναφερθώ καταρχάς ε, στο κατά πόσον το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ορατό, φαίνεται, δραστηριοποιείται και ποιο είναι το μέλλον και οι προοπτικές. Πιστεύω για να βρούμε κατάλληλες ε, λύσεις για το θέμα της ε, δημοσιότητος του ΕΚΤ θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των πολιτικών και εκείνων που λαμβάνουν αποφάσεις και των πολιτών εκείνων που ωφελούνται ή ε, που πρέπει να αποφεληθούν από το Ταμείο. Δυστυχώς πιστεύω ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ ε, των, ε, των εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις και της, του διοικητικού πλαισίου του, της ΕΚΤ και των πολιτών, των δικαιούχων πολιτών Πιστεύω ότι αυτό το χάσμα πρέπει να γεφυρωθεί. Γι' αυτό ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν πάσχει από το να είναι ορατό, ικανοποιητικά ορατό, να φαίνεται δηλαδή ε, πώς ε, λειτουργεί και πώς είναι προσβάσιμο για τους πολίτες μας το, θέμα της ε, δραστηριοποίησης του ΕΚΤ δεν εξαρτάται μόνο από την χρηματοδότηση ε, των ε, των ευρωπαϊκών φορέων αλλά εξαρτάται και από τις παγκόσμιες ανάγκες. Πιστεύω ότι μπορούμε να αυξήσουμε την δραστηριοποίηση του Ταμείου και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της δραστηριοποίησης εθνικών κοινοβουλίων, μέσω εθνικών φορέων, οργανώσεων και αρχών, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοταμείο ε, να γίνει πρώτη λειτουργίας. Πάνω από ένα χρόνο τραβάει η επεξεργασία μιας αίτησης προ το ΕΚΤ. Και αυτό υπό τις καλύτερες συνθήκες. Γι' αυτό πιστεύω ότι το ΕΚΤ από πλευράς ε, λιπτών αποφάσεων θα μπορεί να αυξηθεί η δημοσιότητα, η ορατότητα του Ταμείου αυτού ε, όταν αυξηθεί η αποδοτικότητα της λειτουργίας του πρέπει για να αυξηθεί αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα λειτουργίας ε, πρέπει να στοχεύει σε συγκεκριμένους στόχους. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τη στόχευση των στόχων. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη αριθμητικά στοιχεία. Παραδείγματο χάρη πόσους ε, εργαζόμενους έχει εκπαιδεύσει, πόσοι εργαζόμενοι έχουν καλυφθεί από τα προγράμματα του ΕΚΤ, ε, Πώ επιλέχθηκαν, πόσα προγράμματα έχουν καλυφθεί, πόσα έχουν αρχίσει, πόσες αιτήσει ε, υποβλήθηκαν. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα, απαραίτητα δεδομένα. οι άνθρωποι, οι πολίτες μας πρέπει να καταλάβουν τι κάνει αυτό το κοινωνικό ταμείο, τι έχει επιτύχει, τι προγράμματα έχει, τι επιδιώκει. Οι τελικοί δικαιούχοι, πρέπει να λαμβάνουν εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες. Δηλαδή, ακριβώς η αποδοτικότητα ε, του Ταμείου πρέπει να βελτιωθεί για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα. Οι πολίτες μας αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του ΕΚΤ ως φορέα εξαιρετικής περιπλοκότητας και ότι και αυτό τους αποθαρρύνει, δεδομένου των μακρών διαδικασιών για την έγκριση της αίτησης και την, ε, το ξεκίνημα των προγραμμάτων. Οι πολίτες μας όχι μόνο αποθαρρύνονται, είναι απογοητευμένοι, αλλά θεωρούν και την όλη διαδικασία πολύ ακριβή. Αναγνωρίζω ότι αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις, δεδομένου ότι όλο το σύστημα βασίζεται στην ε, ε, συμμόρφωση και στην τήρηση των περίπλοκων κανόνων λειτουργίας. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με ένα διαφορετικό κουτί εργαλείων, αν θέλετε, με διαφορετικά μέσα. Πρέπει να εισάγουμε νέες ε, αρχές, νέες κατευθυντήριες γραμμές. Για να βελτιώσουμε τις ε, δυνατότητες του Ταμείου χρειαζόμαστε αύξηση του θεσμικού δυναμικού. Το χειρότερο σενάριο που μπορεί να γίνει είναι υπό το βάρος της γραφειοκρατίας και με την πίεση της ε, επιτυχίας σε έργα, σε προγράμματα, να φορτώσουμε άλλο ένα επίπεδο γραφειοκρατικών ελέγχων στο ήδη δυσλειτουργικό ε, κοινωνικό ταμείο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, φτάνουμε στο ΕΤΟΚ. ETUC, η κυρία Τεριάλ, έχει το λόγο αν μπορεί να συντομεύσει λίγο από τα πέντε στα δύο λεπτά. ETUC. Ευχαριστώ. Γαλλικά θα μιλήσω γιατί μπορούμε να το κάνουμε, να μιλήσουμε στη γλώσσα μας. Ε, μου ζητήσατε Εμένα συνδικαλίστρια και γυναίκα ταυτόχρονα μου ζητήσατε να είμαι σύντομη, αλλά εντάξει θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση και θα τα δούμε αυτά λοιπόν. Θα έχετε και την παρέμβαση που θα στώσω γραπτός. Ε, τονίσατε αρκετά σημεία που για μας έχουν ιδιαίτερη σημασία. Πρώτα απ' όλα το πλαίσιο πάνω στο οποίο τοποθετείται, με στο οποίο τοποθετείται αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε από την Επιτροπή για το μέλλον της πολιτικής, της κοινωνικής ε, συνοχής και όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνουμε τι συνεπάγεται αυτό για τη χρηματοδότηση, γιατί ταυτόχρονα έχουμε μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τις δημοσιονομικές προοπτικές μετά από το 2013 και στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων ε, ε, το αναλύουμε αυτό και λέμε όποτε όπως τονίζει η συνθήκη της Αβώνας αυτό που είπε και η κυρία Πρόεδρος για την πολιτική συνοχή ότι θα πρέπει σίγουρα να ενισχυθεί αποτελεί ένα από τους πυλώνες της συνθήκης της Αβώνας εξασφαλίζοντας την ε, αλληλεγγύη ε, στον χώρο και στον τόπο και τον κόσμο ανάμεσα και εκ των πραγμάτων Επιστονίστηκε ο ρόλος του Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού που έχει ενισχυθεί ε, στο έλεγχο, όπως λέμε σε σωστά γαλλικά, το monitoring ε, λογοπαίγνιο της ομιλήτριας για το monitoring, το αγγλικό στα γαλλικά. Λοιπόν, και ακόμα ένα πλαίσιο της σημερινής ε, κρίση οικονομική που διαταράσσει την όλη κατάσταση και το ρόλο με των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα διαχωτικά ταμεία και κυρίως στο κοινωνικό ταμείο το ευρωπαϊκό για να μπορέσει να έρθει μια ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να διδαχθούμε κάτι από τις αποφάσεις αυτές και από τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Επίσης ότι Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στους κανονισμούς και στις προτεραιότητες του Μελλοντικού Κοινωνικού Ταμείου. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, εκεί θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του. Επιβάλλεται κάτι τέτοιο, έτσι. Ε, στον προϋπολογισμό έχει μόνο το 1 τρίτο του προϋπολογισμού στα διευθυντικά ταμεία και να αποτελέσει ένα εργαλείο για τη στρατηγική την ευρωπαϊκή απασχόληση. Και να τονίσουμε ότι μας ανησυχεί αυτό λέω και περισσότερο απλά και μόνο μιλάμε μόνο για μια πρωτοβουλία για την απασχόληση ενώ θα έπρεπε να κάνουμε κάτι περισσότερο για τη στρατηγική αυτή για την απασχόληση και ακόμα για την κοινωνική, για το γενικό χρονοδιάγραμμα, παλιότερα ήταν η πολιτική, κοινωνική, το, το κοινωνικό πολιτικό χρονοδιάγραμμα, που βλέπετε ότι σιγά σιγά απαλήφεται, διαγράφεται, τα τρομερά εμπόδια επίσης σε ένα συντονισμό ενισχυμένο σε διάφορα επίπεδα σίγουρα και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό και τοπικό επίσης επίπεδο. Και στα πλαίσια αυτά Ιδιαίτερα συγκεκριμένα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν ε, για ενέργειες και στο μέλλον και αυτό και για να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και μάλιστα ποιοτική ε, περισσότερε θέσει απασχόλησης και υψηλότερης ποιότητα, επίσης όμως και να ενισχύσουμε την διατήρηση σε εργασίες τους ε, εργαζομένων που θα μπορούσαν να απολυθούν λόγω της κρίσης και που Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει στη Γερμανία μέσα στην, την εργασία, αυτό το Arbeit. Και θα πρέπει, θα πρέπει να διατηρηθούν πάντως τα άτομα αυτά με μια κατάρτιση εκπαίδευση στις θέσεις εργασίας τους. Επίσης, μια καλύτερη συνοχή με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κυρίως όπως επίσης προχωρήσαμε σε βάθος την ανάλυση μας και ξέρουμε ότι όλα αυτά προχωρούν και στο Κοινοβούλιο επίσης για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση που θα πρέπει να ενταχθεί στις μελλοντικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Για ποιο λόγο όλα αυτά συμπληρώνονται με τα μέτρα αυτά ακριβώς του Κοινωνικού Ταμείου που είναι προληπτικής φύσεως ε, για τις συνέπειες ας πούμε για τις μετεγκατάστασης κλπ. Και ενώ αυτά εδώ είναι θεραπευτικά και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων δυστυχώς δεν διασφαλίζεται όπως πρέπει, όπως συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα επανέλθω, είναι αρκετά σημαντικό, είναι οι εταίροι η αρχή αυτή που νομίζουμε ότι είναι κάτι το σημαντικό, η αρχή αυτή να ενισχυθεί, όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά και να ενισχυθεί και να έχουμε ένα σαφή συγκεκριμένο ορισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μην καταφεύγει κανεί μόνο σε εθνικέ πρακτικέ. Εντάξει, ε, να υπάρξει ένα σαφή προσδιορισμό αυτών των εταίρων ε, μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους ε, με ουσιαστικό ρόλο που παίζουν ε, και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τον κοινωνικό διάλογο και επηρεάζει και τη σχέση με την επιχείρηση, με την εταιρεία και ο κοινωνικός διάλογος επίσης θα πρέπει να ισχυθεί. Το προβλέπει ήδη ο σημερινός κανονισμός αλλά δεν έχουν γίνει αρκετά για την υποστήριξη αυτού του κοινωνικού διαλόγου και των κοινωνικών εταίρων, όπως επίσης για την εκπαίδευση και κατάρτισή του, την capacity building, τη δημιουργία προσόντων ακριβώς, αλλά και την ίσχυση όλων αυτών των αποφάσεων στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου και ενεργειών που να χρηματοδοτούνται ακριβώς από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και κάτι ακόμα, πέρα από την εταιρική αυτή σχέση. Νομίζω ότι κανονικά θα ε, ε, οργανωθεί και άλλη ακρόαση πάνω σε αυτό. Θα ήταν κάτι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η νέα και στρατηγική προσέγγιση που την υποστηρίζουμε από τη στιγμή που ε, στενά θα συνδεθούν και οι κοινωνικοί εταιρείε στη λήψη αποφάσεων και στον προορισμό των προτεραιοτήτων και για τα θέματα και περιφερειακά αλλά είμαστε κατά όταν ερχόμαστε σε αυτό το καινούριο, το, αυτό το εξαρτάται που δεν ε, φαίνεται καθαρά ακριβώς τι είναι στις εξηγήσεις που λαμβάνουμε και να δούμε και τι γίνεται με τις κυρώσεις Επίσης τα διορθωτικά ταμεία σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει ε, ένα σεβασμό στο Σύμφωνο Ανάπτυξης και σταθερότητα, γιατί είμαστε και είναι και πολίτες περιφερειών που δεν είναι υπεύθυνοι αυτοί οι ίδιοι για το μη σεβασμό όλων αυτών των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τα κεντρικά όργανα, εθνικά κλπ. Ε, με συγχωρείτε που μακρηγόρησα κάπως. Ευχαριστώ κυρία Λίλια Βολοσνίσκη, Διευθύντρια για θέματα κοινωνικών υποθέσεων και προσπαθήστε σας παρακαλώ να αρκεστείτε στα πέντε λεπτά. Και εγώ στα γαλλικά θα μιλήσω για να είμαι πιο γρήγορο είναι της βιοτεχνίας και των μικρομεσών επιχειρήσεων. Αρκετά πράγματα υπόθηκαν ήδη από τις δύο προηγούμενες ομιλήτριες. Ε, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ. Να επιμείνω όμως σε τρία σημεία την ε, διαχείριση ακριβώς με την αρχή της ε, εταιρική σχέσης, την απλούστευση και το περιεχόμενο, την προσέγγιση το result-based approach, αυτή τη νέα προσέγγιση που έχει να κάνει και με τα αποτελέσματα. Βέβαια, ε, και λυπούμεθα από αυτή η αρχή της εταιρικής σχέσης που κανονικά είναι από τους πυλώνες του Κοινωνικού Ταμείου, όλα αυτά δεν ισχύουν, δεν εφαρμόζονται και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκεί δεν ε, παραπονιόμαστε, αλλά κυρίως σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμμετέχουν αρκετά στις κυβερνήσεις και στις διοικητικές ακριβώς μονάδες, στις τοπικές, για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσο γίνεται περισσότερο το κοινωνικό ταμείο να βλέπουμε καλύτερα τα πράγματα, να είναι πιο αποτελεσματικά, καλύτερη χρησιμοποίηση και απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Γι' αυτό ακριβώ οι κοινωνικοί εταιροί θα πρέπει να συμμετάσχουν σε κάθε επίπεδο, να υπάρχει μια διαχείριση σε κάθε επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώ θα επιθυμούσαμε να υπενθυμίσουμε διάφορε προσπάθειε που πρέπει να καταβληθούν και που στείλαμε αυτέ τι προτάσει στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζουμε ότι συμμεριζόμαστε και από αυτά που λέει εκείνο και τελικά με τη διαχείριση από τι εθνικέ αρχέ για να χρησιμοποιηθούν οι εταίροι αυτοί όσο γίνεται κατάλληλότερα και με ένα, στα πλαίσια ενός μόνιμου διαλόγου και διαρκείς διαδικασίες ανταλλαγών απόψεων και εκεί οι χώρες ε, ε, έχουν προχωρήσει περισσότερο στην ε, χρησιμοποίηση του κοινωνικού ταμείου. Είναι εκεί που συμμετέχουν εταίροι, που είναι κάτι το θεσμοποιημένο. Επίση, μια διαρκή κατάρτιση για ενημέρωση κλπ. ανάμεσα στου ε, υπευθύνου και διάφορε διάφορα μαθήματα και για τις επιχειρήσεις που έχουν δυσκολίες να μπορούν χρησιμοποιήσουν το κοινωνικό ταμείο και που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν, να χρησιμοποιήσουν ακριβώς τα μέσα αυτά ώστε να παραμείνουν στις εργασίες τους εργαζόμενοι εκεί και να αντιμετωπίσουν αυτή τη μετάβαση μέσω μιας ε, διαρκούς ε, κατάρτισης και κατάλληλη πολιτική στην αγορά εργασίας. Εδώ στο κοινωνικό αυτό ταμείο το 5-3 άρθρο μιλά για την ενίσχυση αυτών των των δυνατοτήτων των ε, κοινωνικών εταίρων και το άρθρο αυτό ακριβώς συντάχθηκε για να υποστηρίξει την δημιουργία ε, αυτών των δυνατοτήτων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ε, θα θέλαμε να ισχύσει αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί οι οργανώσεις, οι κοινωνικοί εταίροι για τη βιοτεχνία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν ήδη τη δυνατότητα από μόνο της να είναι ενεργά αναμειγμένοι στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Θα θέλαμε το άρθρο αυτό να μην περιορίζεται μόνο στα κράτη-μέλη τα νέα από τα ιδιαίτερα προβλήματα και κριτική που είχε ασχεθεί στο Ευρωπαϊκό Ενεργό Ταμείο είναι ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Σχετικά με τη διαδικασία του υπάρχει μια καμψία, μπορούμε να πούμε, στην οικονομική διαχείριση. Γι' αυτό ακριβώ επιγόντω χρειάζεται να ενισχύσουμε την απλούστευση και σε διοικητικό επίπεδο ε, και οργανωτικά. Και εκεί υπάρχουν διάφορε προτάσει μέσω τη γενική ενίσχυση και επίση τη δυνατότητα να έχουμε διάφορε μεταφορέ ανάμεσα στι προτεραιότητε, στα επιχειρήματα επιχειρησιακά προγράμματα και επίσης να μπορέσουν να ισχύσουν να βαντεμεκούμ μια βέλτιστη πρακτική ακριβώς για τις υποχρεώσεις, πώς είναι τα, τα πράγματα να απλοποιηθούν και επίσης τη σύσταση τεχνικών ομάδων για τη διαχείριση όλων αυτών των ε, θεμάτων, των ε, σχεδίων και οικονομική, από οικονομικής πλευράς για να δούμε ακριβώς, να εξετάσουμε αναλυτικότερα αυτές τις δικές διαδικασίες και να τις απλοποιηθεύσουμε. Επίσης, όσον το περιεχόμενο, είμαστε υπέρ του FSA που θα πρέπει να υποστηρίξει την πολιτική της Ένωσης για το 2020 και επίσης αυτή η, FXB, η Flex Security ε, που να πρέπει να υποστηριχθεί πλήρως, δηλαδή να λεφθούν υπόψη τα προβλήματα της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, επίσης διαρκούς κατάρτισης, διαβίου κατάρτισης, όπως επίσης και ενεργές πολιτικές στην αγορά εργασίας. Και υποστηρίζουμε πάντα αυτή τη νέα προσέγγιση, το result-based approach, ε, και επίσης ε, μια ριζοσπαστική αλλαγή αντίληψης σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις. Απαιτείται αυτό για να ισχύσουν όλα αυτά. Χρειάζονται προσαρμογές κατάλληλες και κυρίως με τα μέτρα να δούμε πώς θα επηρεάσει το FSA αυτό την αγορά εργασίας και ακριβώς τις δυνατότητες για να ξεφύγει κανείς από τη φτώχεια. Εντάξει, έχω ακόμα λίγο για να μιλήσω και επίσης ε, να δούμε όσοι διαχειρίζονται αυτά τα προγράμματα και τα μέτρα κατάρτισης για αυτούς που κάνουν την ε, ανάλυση τους και όσους αναλύουν αυτά τα προγράμματα ακριβώς. Εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε το χρόνο σας. Τώρα ερχόμαστε στη CRPM, τη Συνομοσπονδία των θαλάσσιων περιοχών. Έχουμε την κυρία Μαριάνο και την κυρία Μπεσίλ. Δεν ξέρω πώς θα τα κατανείματε μεταξύ σας. Έχετε πέντε λεπτά να μοιράσετε. Ευχαριστώ. Δεν θα μακρηγορήσουμε. Θα ήθελα απλώ να σας εξηγήσω τι είναι αυτή η διάσκεψη περιφερειακών ε, θαλασσίων περιοχών. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μας καλέσατε σήμερα εδώ, στην ακρόση αυτή σε, σε αυτό το θα έλεγα καθαρά γυναικείο πάνελ. Η CPMR ε, εκπροσωπεί 160 περιφέρειες ε, στην Ευρώπη και όλες αυτές οι περιοχές ε, ε, εμπίπτουν σε ένα ε, πλαίσιο κοινωνικής συνοχής και στο πέμπτο πρόγραμμα πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής. Βεβαίως έχουμε μέσα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής άμεση επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μία από τις ομάδες εργασίας του CPMR εργάζεται βασικά για εργασιακά θέματα, λειτουργεί, ε, επικεντρώνεται κυρίως σε εργασιακά θέματα και θα δώσω το λόγο στην κυρία Κατρίν Βεσί, η οποία είναι η αντιπρόεδρος της περιφέρειας της Ακιτέν, για να σας εξηγήσει την εργασία της. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι οι περιφέρειες υποστηρίζουν το ΕΚΤ σαν εργαλείο περιφερειακής πολιτικής για συνοχή στην Ευρώπη. Έχουμε μια πολυδιάστατη κρίση και βεβαίως πρέπει να μειώσουμε τα τεράστια χάσματα που υπάρχουν μεταξύ των διαθέσιμων προσόντων και των απαιτούμενων προσόντων της αγοράς εργασίας. Είναι θέμα προσβασιμότητας στην απασχόληση ορισμένων κοινών που κινδυνεύουν να αποκλειστούν. Είναι δύσκολο να περιγράψουμε το πλαίσιο. Υποστηρίζουμε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της στρατηγικής για το 2020, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Στην CRPM αναλύσαμε αυτά που προτείνονται στη στρατηγική του 2020 και συζητήσαμε με την κυρία Πασκάλ Πρένη που ήταν η μόνιμη εισηγήτρια για το, για το ΕΚΤ. Οι περιφέρειές μας ήδη εφαρμόζουν τις προτάσεις και ήδη έχουν την υποστήριξη την ενεργή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Επιμένουμε λοιπόν ότι αυτό το ταμείο είναι πολύ σημαντικό για μας, εδαφικά μάλιστα. Έχει, ο ρόλος του είναι σαφής, πρέπει να συμβάλλει στην σε μια ανάπτυξη που να περιλαμβάνει όλους, ιδιαίτερα για την απασχόληση και ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν ανάγκη κατάρτισης. Οι προηγούμενοι παρεμβαίνοντες ακριβώς τόνισαν ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτούς που έχουν απομακρυνθεί περισσότερο από τα απαιτούμενα προσόντα για την αγορά εργασίας και έχουν ανάγκη κατάρτισης για να μην βρεθούν εκτός επιχειρήσεων. Για να εφαρμόσουμε αυτή την αποστολή ε, πρέπει να βρούμε μία απάντηση από τις, τις διάφορες περιοχές. Δηλαδή πρέπει να μπορέσουν οι άνθρωποι να μείνουν στις περιοχές τους με αξιοπρέπεια και να εργαστούν. Γι' αυτό το λόγο υποστηρίζουμε τις προτάσεις της Επιτροπής, της Κομισιόν, που περιλαμβάνονται στην πέμπτη έκθεση συνοχής, ειδικότερα δε τις προτάσεις που προ, ε, προτείνουν ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο το οποίο θα αναλυθεί στα κράτη-μέλη μέσω συμβάσεων εταιρικής σχέσης. Αυτές οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης πρέπει να προετοιμαστούν με τις περιφέρειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πρόκληση. Θα θέλαμε λοιπόν όλα αυτά να συνεχίσουν μέσα στο περιφερειακό πλαίσιο ώστε να ομοδοποιηθούν τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά εργαλεία. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σημεριζόμαστε την ανησυχία να μειωθεί ε, η επιρροή του ΕΚΤ. Πιστεύουμε ότι το ΕΚΤ και το ΦΕΔΕΡ πρέπει από κοινού να ενεργήσουν και γι' αυτό χρειαζόμαστε συμπληρωματικότητα μεταξύ τους. Ακόμη η αποτελεσματικότητα του ΕΚΤ ε, συνεπάγεται επικέντρωση στα αποτελέσματα και πρέπει να δούμε αν πραγματικά έχουμε υλοποιήσει τον στόχο μας όταν κινητοποιούμε κονδύλια στα διάφορα ε, εδάφη. Δηλαδή τελικά προετοιμάσαμε καλύτερα τους πληθυσμούς μας, τους πιο εύθραυστους για να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Αυτή είναι η ερώτηση. Όλα αυτά βεβαίω απαιτούν και απλούστευση του ΕΚΤ. Θα υπάρξουν και προτάσεις εκ μέρους μας σε σχέση με την απλούστευση που απαιτείται. Πιστεύουμε δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχουν σταθεροί και απλοί κανόνες για τη χρηματοδότηση. Τέλος, ως προς τη διακυβέρνηση από τους εταίρους, ε, έχουμε κάνει κάποιες αναλύσεις και πρέπει να σας πω ότι οι περιφέρειες ήδη εφαρμόζουν τις προτεραιότητες του 2020 και αυτό μέσα στο ένα πλαίσιο κάθε της ε, διακυβέρνησης αλλά και οριζόντιας με όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους. Η ανάπτυξη στρατηγικών για την απασχόληση περιφερειακά περνάει από τη δέσμευση των επιχειρήσεων, των οργανώσεων και των ενώσεων. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να δικτυωθούν εδαφικά για να καλύψουν την απασχόληση. Και θεωρούμε ότι το ΕΚΤ λοιπόν είναι ένα σημαντικό εργαλείο για το μέλλον μέσω των λύσεων που θα προτείνει στα διάφορα εδάφη και πληθυσμούς ώστε να αποσβέσουμε ε, να αποδυναμώσουμε μάλλον τις επιπτώσεις της κρίσης που δυστυχώς δεν έχει ακόμη τελειώσει. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο κύριος Κονιγόητο έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επιτροπή Απασχόλησης που μας κάλεσε. Θα μιλήσω αγγλικά. Η κοινωνική πλατφόρμα εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών και δεν εκπροσωπούμε τους κοινωνικούς εταίρους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μας δείτε από διαφορετική οπτική γωνία, από τους κοινωνικούς εταίρους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το θέμα είναι, εμείς αναρωτιόμαστε ποιο είναι το νόημα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δεδομένου ότι ζούμε σε εποχές λιτότητας, σε, σε εποχές δύσκολες. Η πραγματικότητα στην αγορά εργασίας είναι, δείχνει δυστυχώς ότι δεν ακολουθεί τις, αισιόδοξε τις προοπτικές για οικονομική ανάκαμψη. Η Ίγκε Μετάλλη, το μεγαλύτερο συνδικάτο στη Γερμανία, είπε ότι 45% των μελών της έχει μερική απασχόληση ή συμβάσεις εργασίας για μικρό χρονικό διάστημα και μόνο 15% έχουν πλήρη απασχόληση της συνδικαλιστικής αυτής ένωσης. Ποιο είναι λοιπόν το μέλλον, ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Σίγουρα δεν θα είναι όπως τις περιγράφει το κοινωνικό ταμείο. Άρα λοιπόν αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο σκοπός λειτουργίας αυτού του ταμείου. Είναι για να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει τα κονδύλια τα οποία περικόπτουν τα κράτη-μέλη. Δηλαδή θα χρηματοδοτεί τα κενά ή για να θα επανέλθουμε σε κάτι το οποίο έχει ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του τέστην την ενεργό πολιτική ενσωμάτωσης που ήταν και η πρώτη μας απέτηση για τη δημιουργία του Κοινωνικού Ταμείου. Πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε τι είδου συνοχή και πώς θα εφαρμόσουμε τη συνοχή στο πλαίσιο του, του 2020. Τι είδου ευέλικτα προγρήματα θα εφαρμόσουμε για την αγορά εργασίας. Τι θα γίνει για τη σχέση μεταξύ του ΕΚΤ των πιστώσεων και τις προοπτικές για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Τι εννοούμε με νέες δεξιότητες, είναι μόνο νέες τεχνολογίες, είναι μόνο, αφορά μόνο τους ανθρώπους που έχουν ήδη ψηλά προσόντα ή στοχεύει σε ανθρώπους που έχουν χαμηλά προσόντα. Παραδείγματο χάρη στη Γαλλία καλύπτει το επίπεδο 6. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιου ανθρώπους καλύπτει με ποια προσόντα το ΕΚΤ. Επίσης επανέρχεται και ε, ε, παλιές συζητήσεις, η συζήτηση του Λόκνες για την ε, διευκόλυνση της, της κινητικότητας Ήμουν ε, απελπισμένος όταν είχαμε τη συζήτηση αυτή για τη γραφειοκρατία και το διοικητικό άχθος. Με 15 χρόνια αργότερα έχουμε ακόμα τεράστια γραφειοκρατία και διοικητικό βάρος. Έχουμε λοιπόν σαφώς ένα πρόβλημα στην διοίκηση, στο διοικητικό μέρος. Έχουμε ένα πρόβλημα του ταμείου δηλαδή στο χρηματοδοτικό μέρος και σαφώς ένα πρόβλημα ε, στην, ε, στους στόχους Ποιο, ποιος είναι ο στόχος της συγχρηματοδότησης. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία λόγω των οικονομικών δυσκολιών δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα συγχρηματοδότησης. Έχουμε επίσης και μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και εμπίπτουν και αυτές στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης. Πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε ποιος μπορεί και τι μπορεί να κάνει στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης. Άρα αυτή τη στιγμή προκύπτει το ερώτημα τι επιδιώκει το Ταμείο, ποιο, ποια κατάρτιση, ε, ποιοι, ποιοι εργαζόμενοι θα καλυφθούν με ποιο είδους κατάρτισης και απόκτηση δεξιοτήτων και πρέπει επίσης να διευκρινίσουμε τι μέσα, τι εργαλεία πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα, τα κράτη-μέλη για να εκτελέσουν τα προγράμματα και ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ του κοινωνικού φόρουμ και των κοινωνικών εταίρων. Πρέπει να σας πω ότι εμείς ε, ως μέλη της κοινωνικής πλατφόρμας είμαστε εκτός των συζητήσεων που γίνονται με τους κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτουν οι συζητήσεις, να ενσωματώνουν και την κοινωνία των πολιτών. Και τέλος πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση που να επικεντρώνεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα μας ενδιαφέρουν. Δεν πρέπει να έχουμε μόνο στα κατά νου τις στατιστικές. Εμείς δεν στοχεύουμε μόνο σε ποσότητα, σε δεδομένα. Θέλουμε και ποιότητα. Θέλουμε να ε, προσφέρουμε ποιότητα η οποία να μπορεί να προωθήσει της απόκτηση νέων δεξιοτήτων στις νέες θέσεις εργασίας. Ήπιες ε, μορφές απασχόλησης απασχόλησης και διαπολιτισμικές μορφές απασχόλησης. Ποιότητα λοιπόν, μην το ξεχνάμε αυτό. Και Είμαστε εντελώς αντίθετοι στη χρησιμοποίηση των ε, πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου ως μέσον επιβολής κυρώσεων σε κράτη-μέλη τα οποία δεν μπορούν να ε, καλύψουν τις υποχρεώσεις τους λόγω της οικονομικής κατάστασης και να χρησιμοποιηθεί ως μέσον ε, κυρώσεως για την αγορά εργασίας. Είμαστε λοιπόν αντίθετοι με τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων για κυρώσεις και ποινές. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε το μέλλον του ΕΚΤ. Βεβαίω έχουν να παίξουν ρόλο οι κοινωνικοί εταίροι, αλλά οπωσδήποτε ε, και οι κοινωνικές οργανώσεις και φορείς πρέπει να παίξουν ένα ρόλο, διότι εμείς γνωρίζουμε, είμαστε στην πρώτη γραμμή που υπάρχουν συγκεκριμένε ανάγκες. Σας ευχαριστώ που δώσατε το λόγο και ε, λίγο που ξεπέρασα το χρόνο εργασίας μου. Ε, Σας ευχαριστώ. Ε, σύντομα για να μπορέσουμε να έχουμε μια συζήτηση. Η κυρία Λέσκα και μετά η κυρία Σρέντερ. Dziękuję Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο Ελίζαμπεθ για την προετοιμασία αυτής της ακρόασης και για την πρόσκληση ε, εμπειρογνωμόνων ε, από διάφορους τομείς που μπορούν να μας πούν ποιες είναι οι εμπειρίες τους για τη χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και ευχαριστώ όσοι έλαβαν το λόγο για τα πολύ ενδιαφέροντα μα είπαν, αλλά ορισμένα σημαντικά έλειπαν, στοιχεία σημαντικά που έχουν πραγματικά σημασία. Μιλήσατε, είπατε ότι περισσότερη αποτελεσματικότητα στη χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού αμείου, αλλά δεν ακούσαμε καμία πληροφορία και καμία δήλωση στι εισηγήσει σα που να λένε ότι αυτή η χρησιμοποίηση θα πρέπει να συνδέεται άμεσα και με τον έλεγχο των αναγκών της αγοράς εργασία. Θα πρέπει να σας πω κάτι, ότι και στο παρελθόν είχα την ευκαιρία να, να ζήσω κάτι το τρομερά σημαντικό και από τους Δανούς και άλλους ε, έμαθα πολλά πράγματα για την αγορά εργασίας, για την οργάνωση, για τα προσόντα των εργαζομένων, όλα αυτά πώς συνδυάζονται και συνδυάζονται με την αγορά εργασίας. Και νομίζω ότι αποτελεί από τα στοιχεία τα πιο αδύναμα, τους αδύναμους κρίκους, τη χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και θεωρώ ότι θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε εδώ λύσεις ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή. Πριν από μερικές εβδομάδες μου ζήτησαν κάτι, συμβουλές δηλαδή και συστάσεις σχετικά με το συνδυασμό αυτό και μιλάω για την δική μου περιφέρεια από την Πολωνία, μια περιοχή που ηγείται στην, ε, είναι μπροστά στη χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και μου ζήτησαν να δημιουργήσω μια πλατφόρμα, ας την πούμε έτσι, κάτι για να προετοιμάσει τους φοιτητές, τους σπουδαστές φοιτητές για να μπορέσουν να βρουν δουλειά μετά στι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι, μια οργάνωση, μια κατάλληλη δομή για την προετοιμασία των ε, μελλοντικών ε, ε, τελειοφύτων που θα μπορέσουν επαναλαμβάνω να εργαστούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και στα πλαίσια αυτής της οργάνωσης και δομής θα μπορούσαμε να έχουμε εκπαιδευτές που να γνωρίζουν κατάλληλα ποιε είναι οι ανάγκες των διαφόρων επιχειρήσεων, όσους προλαμβάνουν προσωπικό στις διάφορες επιχειρήσει και να προετοιμάζουν τους σπουδαστέ ώστε από τη στιγμή που θα έχουν το δίπλωμά τους ε, να μπορούν να εργαστούν άμεσα και να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για να βρουν δουλειά και επίσης για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης επαναλαμβάνω, και την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξης να σας πω ότι εδώ τα πράγματα είναι κάπως απλά γιατί εκεί όλα αυτά συνδυάζονται με τα διαφορά σχέδια ανάλογα με την όλη οργάνωση και εμείς θα πρέπει ε, νομίζω ότι για να αλλάξουμε την αντίληψη του κόσμου πάνω στη χώρα μου να συντάξουμε ένα σχέδιο, να το συντάξουμε κατάλληλα και να μπορέσουμε μετά να χρηματοδοτηθούμε και χρηματοδότηση προκαταρτική ακριβώ για να το συντάξουμε, να το προχωρήσουμε αυτό το σχέδιο. Από τη στιγμή που θα έχουμε τα χρήματα αυτά, προχωράει το σχέδιο πάρα πολύ γρήγορα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και εδώ η κατάσταση να σας πω ότι εδώ πια είναι πολύ διαφορετική. Στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συντάσσεται πρώτα ένα σχέδιο, μετά δίδονται τα χρήματα γίνεται συμφωνία και τότε μόνο βλέπουμε ποιοι θα είναι οι τελικοί αποδέκτες που θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου. Όλα αυτά δεν είναι και τόσο αποτελεσματικά πάντα, γιατί αυτοί οι αποδέκτε δεν συμμετέχουν πάντα σε κάτι το οποίο πραγματικά να χρειάζονται. Έχουμε και διάφορα ακραία εντελώ παραδείγματα και στη χώρα μου, την Πολωνία και αλλού. Δηλαδή, πώ θα μπορέσουμε να ελκύσουμε αυτού του αποδέκτε, του τελικού. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μα δείχνουν ότι εκείνοι που τελικά υποφελούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι οι επιχειρήσει οι οποίε προσφέρουν κατάρτιση και όχι οι ίδιοι τελικοί αποδέκτε, έτσι οι τελικοί χρήστε. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να το συλλογιστούμε δούμε αυτό σαν πρόβλημα. Και επίσης ε, πώς θα δίδονται τα κονδύλια αυτά στα πλαίσια ενός σχεδίου, ενός προγράμματος, γιατί βλέπουμε ότι το 25% των κονδυλίων μπορεί να πάνε στη διοίκηση, αλλά μόνο το 10% για την αγορά ας πούμε υλικού. Και θεωρώ ότι η αναλογία αυτή θα πρέπει να αλλάξει για τη χρήση των κονδυλίων. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Επίσης θα ήθελα να ξέρω, να μου πείτε πώς, ε, τι θα, ποια άποψη έχουν οι συγκεκριτές. Ναι, θα μπορούσατε να ρωτήσετε από τους ομιλητές ορισμένα πράγματα. Θα έχουμε έτσι κι ε, ανάμεσά μας πολλέ πολλές άλλες ε, φορές να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα και τους προστατευσμού και την απόψή μας για το μέλλον. Αλλά σήμερα θα πρέπει να υποβάλουμε ερωτήσεις, επαναλαμβάνω, στους ε, και συγγήτριες Σρέτερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συμμετέχοντες, όσοι ήρθαν εδώ, παρόλο που μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, πιστεύω ότι και οι γραπτές συνεισφορές είναι πολύ χρήσιμες. Έχουμε δύσκολο έργο μπροστά μας. Θα αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα. Καταρχάς πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που θέτεται στο επίκεντρο την ε, συμμετοχή, την, την, εταιρική συμμετοχή και την ε, συνεργασία μεταξύ των εταίρων. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά ε, παραδείγματα όπου αυτή η συμμετοχική πλατφόρμα έχει μεταφραστεί σε, σε πράξη, σε έργα και με οικονομική υποστήριξη. Όμως ε, υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα παραδείγματα όπου απέτυχε αυτή η συμμετοχική διαδικασία, αυτή η συνεργασία. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε τα κράτη-μέλη εκεί όπου δεν πέτυχαν αυτά τα προγράμματα να καταβάλουν καλύτερες προσπάθειες. Αυτή λοιπόν η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει περιθώριο βελτίωσης. Στην ε, προετοιμασία τώρα του νέου προϋπολογισμού μπορούμε να προβλέψουμε μέτρα ε, ανάπτυξης των πρωτοβουλειών αυτών ε, για το επόμενο έτος. Τώρα, πώς θα καθορίσουμε, πώς θα χειριστούμε το θέμα του ενιαίου ορισμού. Ε, αυτό θα δούμε πώς θα γίνει. Πρέπει να ε, εφαρμόσουμε μέτρα αποκέντρωσης, τα οποία δεν θα περιορίσουν την ευελιξία εάν έχουμε νέα, νέους στόχους, νέα προγράμματα στο ΕΚΤ και βεβαίως θα έχουμε καινούργια προγράμματα και καινούριου στόχους, διότι αυτή, αυτό είναι το καινούριο στοιχείο με την προοπτική του 2020, οι αλλαγές αυτές. Δεν μπορέσαμε να περάσουμε αυτές τις αλλαγές και τις πρωτοβουλίες που επισημούσαμε στο παρελθόν. Τώρα όμως ε, δεδομένου ότι εστιάζουμε την προσοχή μας ιδιαίτερα στην ανταγωνιστικότητα, θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε αυτές τις ε, σημαντικές αλλαγές. Τι σημαίνει αυτό τώρα μέσα στο πλαίσιο των, της συνεργασίας. Χρειαζόμαστε καινούριου συνεργάτες. Τι πιστεύετε εσείς, ποιοι άλλοι συνεργάτες πρέπει να καλυφθούν από το ΕΚΤ. Ε, να το δούμε από μια πανευρωπαϊκή σκοπιά και όχι από εθνική σκοπιά εν συνεχεία όσον αφορά το θέμα της, ε, ε, του conditionality έχει η Κομισιόν τρεις στόχους που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστοί. Τα κράτη-μέλη να θέσουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις όσον αφορά την διάθρωση της νομοθεσία τους και για να δούνε, να η ευκαιρία λοιπόν να εξετάσουν αν έχουν ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για να εφαρμόσουν αυτές τις ε, νέες δομές. Επίσης ε, έχετε αναφέρει και το Global Grant, το οποίο βεβαίως υφίσταται αλλά δεν εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις η, στη δεύτερη σειρά των κανονισμών που θα εξετάσουμε χρησιμοποιείται αυτό το Παγκόσμιο Ταμείο αλλά δεν χρησιμοποιείται συχνά. Πώς είναι δυνατό να πείσουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσον. Διότι ορισμένα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτές τις πιστώσεις, ε, αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα με εξαιρετική επιτυχία με εκπλήττει το γεγονός ότι δεν άκουσα καμία πρόταση για βελτίωση της λειτουργίας του Global Grant, αυτού του παγκόσμιου, της, ενίσχυσης με, παγκόσμια προοπτική. Θα ήθελα λοιπόν, ε, και δεδομένου ότι αυτό θα μας απασχολεί στο μέλλον, να ακούσω τις απόψεις σας. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις ομιλίες, τις εισηγήσεις. Στην κρίση αυτή που διανύουμε, το ΕΚΤ βεβαίως ε, χρησιμοποιήθηκε αποτελεσματικά για να μην χειροτερεύσει περισσότερο η αγορά εργασίας και για να βοηθήσει όσο το δυνατόν μια κοινωνική, το στοιχείο της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Αυτά πρέπει να τα διατηρήσουμε στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Ε, θα ήθελα να ακούσω ε, πόσο σε ευρωπαϊκή διάσταση μπορεί το ΕΚΤ να υποστηρίξει προτεραιότητες ε, δικές μας. Όταν εργαζόμαστε στο, στο, επί του μέσου διευκόλυνσης μικροεπενδύσεων και επενδύσεων, ε, χρηματοδοτικών επενδύσεων μικρής εμβέλειας ε, είχαμε συζητήσει πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους μικρούς επιχειρηματίες ε, και να τους παρακολουθήσουμε, να τους εποπτεύσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό το μέσα στο πλαίσιο της μικροχρηματοδότησης επιχειρηματιών. Και επίσης, άλλο θέμα, όταν μιλάμε για την διαβίου εκπαίδευση, κατάρτιση, απόξη δεξιοτήτων διαβίου, αυτό το πλαίσιο δηλαδή, εάν λάβουμε υπόψη τις ε, ανάγκες ανάπτυξης στην παιδική ηλικία και την ανάγκη ε, εκπαίδευσης παιδιών από, μειονεκτικά, ε, από μειονεκτικό κοινωνικό περιβάλλον ή κοινωνικό περιβάλλον, ε, εδώ πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες εδώ να χρηματοδοτηθούν προγράμματα, να διαμορφωθεί μια στρατηγική από το ΕΚΤ για την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιδιών ήδη στη σχολική, μαθητών δηλαδή, σχολική ηλικία, Διότι αν λάβουν αυτά τα εφόδια θα μπορέσουν να είναι αργότερα επιτυχείς ε, στην αγορά εργασίας, καλοί εργαζόμενοι. Επίσης η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Ρωμά ε, θα ήθελα να ξέρω πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα. Έχουμε ε, συζητήσει επιμακρών για αυτό το θέμα στο Κοινοβούλιο με διάφορα μέτρα και ψηφίσματα. Η κυρία Μπάουερ, μετά η κυρία Τσίμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι πληροφορίες που μας... και ευχαριστώ όλες τις ομιλήτριες μέχρι τώρα και ομιλητή ε, για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσαν. Ιδίω τώρα που πρέπει να εργαστούμε ε, πάνω σε μια καινούρια έκθεση, νέο πρόγραμμα που αφορά το δυναμικό απορρόφησης. Ακούσαμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στην απορρόφηση των πιστώσεων, των κονδυλίων. Συμβαίνει λοιπόν το εξής. Οι ενισχύσεις και η στήριξη δεν φτάνει στους, πολλές φορές τους δικαιούχους που κατοικούν παραδείγματο χάρη σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε ε, πολύ μικρές περιφέρειες δεν λαμβάνω, λοιπόν την ενίσχυση και τη βοήθεια που πρέπει. Ρωτώ λοιπόν το εξής. Ποιε ευκαιρίε μας προσφέρονται για να αυξήσουμε το δυναμικό απορρόφησης των πιστώσεων. Η κυρία Τσίμερ. Ευχαριστώ για τις εισηγήσεις και τα σχόλια. Θα είμαι πολύ σύντομη δεδομένου ότι Συμφωνώ με πολλούς από τους προλαλήσαντες. Μέχρι τώρα αυτά που ακούσαμε έδειξαν ότι περισσότερα ερωτήματα τίθενται από ότι ε, προβλήματα τα οποία έχουν λυθεί. Όλο και καινούργια προβλήματα, ζητήματα προκύπτουν. Αυτό το οποίο Επισημένο είναι ότι μέχρι τώρα όσοι μίλησαν εκπροσωπούν στενά ε, την οργάνωση ή τον φορέων από τον οποίο στάλισαν εδώ. Ε, εγώ θα ήθελα να δω μία αντιμετώπιση πιο ευρεία, ε, δεδομένου ότι μιλάμε συνέχεια για το πλαίσιο συνεργασίας, το συνεργασίας μεταξύ των εταίρων. Άρα, λοιπόν, για τα διορθωτικά ταμεία, για το Ταμείο Συνοχής, ε, πρέπει να δούμε μια κοινωνική προοπτική, ε, όχι ο καθένας στα στεγανά της οργανώσεως και του φορέα του να εκφράζει τις απόψεις του και να ζητά το α και το β. Πρέπει οι στόχοι μας να είναι πιο ευέλικτοι και ευρύτεροι ε, και τα αιτήματά μας προς το ΕΚΤ πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να εξηγήσουμε στους ενδιαφερόμενους τι εννοούμε, ποιος είναι ο ρόλος πώς, μπορεί ε, το ΕΚΤ να μεταβάλει ε, ε, τη, τα προγράμματά του, να εφαρμόσει τα προγράμματά του στην πραγματικότητα και πώς μπορούν όλες αυτές οι αιτήσει να μεταβληθούν σε έργα. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να προσαρμόσουμε το Ταμείο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας εάν, αλλά θα πρέπει και οι ενδιαφερόμενοι φορείς να προβάλλουν τα αιτήματά τους προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας ε, και, και ιδίω σε μικρότερα προγράμματα, μικρού εύρους. Διότι διαφορετικά, αν ο καθένας προβάλλει αιτήματα μόνο για το συγκεκριμένο του φορέα ή οργανισμό, δεν θα επιτύχουμε την κοινωνική ενσωμάτωση. ε, όσον αφορά τους στόχους για την καταπολέμηση της φτώχειας της Ευρώπης 2020, πάρα πολλοί πιστεύουν, όπως οι εκπρόσωποι του ΕΠΣΚΟ, ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Δεν είναι εφικτοί οι στόχοι που αφορούν την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ατζέντα 2020. Τι λοιπόν πρέπει να γίνει αν από τώρα εκφράζονται αυτές οι επιφυλάξεις. Ευχαριστώ. Έχω μια ευρύτερη ερώτηση, δεν απευθύνεται σε κανένα ειδικότερα. Αλλά στις συζητήσεις που έχουμε εδώ και καιρό εμπλέκονται διάφορες προσεγγίσεις. Το ερώτημα συνεπώς είναι ότι ε, πρέπει το Ταμείο να έχει μια αυτονομία περιφερειακή ή πρέπει τελικά όλα τα πράγματα να είναι πολύ επισημασμένα όσον αφορά τη στρατηγική του 2020. Άλλο ερώτημα που έχω στο μυαλό μου είναι ο βαθμός αυτονομίας σε σχέση με το ΦΕΝΤΕΡ. Δηλαδή, πρέπει να διατηρηθεί αυτή η πλήρης αυτονομία ή οι περιφέρειες πρέπει να έχουν ένα συνολικό φάκελο με τον οποίο να διαχειρίζονται και τα δύο ταμεία, τα κονδύλια και από τα δύο ταμεία. Τρίτη σκέψη, αναφέρθηκατε και εσείς στα σχόλιά σας, είναι η σπουδαιότητα που πρέπει να αποδοθεί στην διασύνδεση με τους κοινωνικούς εταίρους. Πώς βλέπετε δηλαδή το σημερινό μηχανισμό, ε, τι πρέπει να βελτιωθεί. Αντιλαμβάνομαι όσα προκύπτουν από τις ε, ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Αλλά υπάρχουν και από την άλλη πλευρά οι εθνικές, τα εθνικά εμπόδια. Και ε, κανείς πρέπει να μπορεί να διακρίνει που πρέπει να απευθύνει την απέτησή του, το αίτημά του. Άλλο θέμα πάλι που μας απασχολεί είναι τα αποτελέσματα του ΕΚΤ. Όλοι είπατε ότι πρέπει να είναι ε, λιγότερο γραφειοκρατικό κτλ. Σύμφωνοι. Αλλά σύμφωνα με εσά, ποια είναι η σωστή αξιολόγηση όσον αφορά την μεθοδολογία. Δηλαδή τελικά τι αξιολογούμε, τον αριθμό των θέσεων εργασίας ε, που δημιουργήθηκαν, ε, τον αριθμό των χαμόγελων στην περιοχή, ε, τι αξιολογούμε δηλαδή. Εντάξει υπάρχει η αξιολόγηση για να ικανοποιείται το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά ε, πρέπει να έχουμε και την αξιολόγηση των δικαιούχων. Ένα άλλο θέμα είναι το εξής. Αν συμφωνήσουμε και πούμε ότι μέχρι το 2020 δεν θα έχουμε αρκετά κονδύλια, οπότε πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τα μέσα εφαρμογής της στρατηγικής. Αυτό σημαίνει άραγε ότι πρέπει να μεταβάλουμε τις προτεραιότητες μέσα στο ΕΚΤ. Δηλαδή, από τι καταλαβαίνω, υπάρχει μία συζήτηση για το κατά πόσο η απασχολησιμότητα επαρκεί ή αν πρέπει να ενισχύσουμε την καταπολέμηση της φτώχειας και ενδεχομένως τότε να χρειαζόμαστε παρέμβαση του ΕΚΤ περισσότερο ανάντι συμπεριλαμβανομένης και της καταπολέμησης του αποκλεισμού. Ένα άλλο θέμα και ομολογώ ε, πολλά, πολλές είναι οι ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα γύρω από αυτό το ενδιαφέρον θέμα που έχουμε σήμερα. Ε, ένα άλλο θέμα έχει περισσότερο σχέση με το Φεντέρ, όχι αποκλειστικά. Ε, το σχόλιο της κυρίας Γιαζεύσκα. Συχνά έχουμε την εντύπωση ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία στην πραγματικότητα ενεργοποιούν κυκλώματα οικονομικά και δίκτυα τα οποία ευνοούν τα άλλα κράτη-μέλη. Αναφερθήκατε στις υποδομές. Ε, Βεβαίω αυτό συσχετίζεται περισσότερο με το φετέρ μέσα στο πλαίσιο του ΦΕΝΤΕΡ έχουμε μια αυτοκινητόδρομο ή μια γέφυρα που θα κατασκευαστεί σε μια χώρα και είναι επιλέξιμο και από την άλλη πλευρά οι εταιρείε ε, που θα υλοποιήσουν αυτό το έργο υποδομής προέρχονται από όλες τις χώρες ε, και δεν χρειάζονται τα λεφτά του ΦΕΝΤΕΡ. Ε, Αντιμετωπίζετε το ίδιο πρόβλημα με το ΕΚΤ ή όχι. Η κυρία Μωρά νομίζω έχει και αυτή ερωτήσεις και μετά θα απαντήσετε όλοι. Ε, και θα έχετε λίγο χρόνο βεβαίως. Ε, ε, δεν θα προσθέσω πολλές ερωτήσεις, λέει η κυρία Μωράν, γιατί τελικά οι απαντήσεις μας ενδιαφέρουν, γιατί έχει περάσει και ο χρόνος. Ένα θέμα θέλω να προσθέσω, πολύ σημαντικό. Τι διασύνδεση υπάρχει μεταξύ ευρωπαϊκής πολιτικής, εθνικής πολιτικής και τοπικής πολιτικής όσον αφορά την απασχόληση. Δηλαδή, πώς μέσω του ΕΚΤ μπορούμε να εξασφαλίσουμε την συνέπεια μεταξύ αυτών των τριών επιπέδων πολιτικής και στόχων. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν με την ίδια σειρά. Η, η κυρία Μαρζένα Τσιλιεύσκα λοιπόν, έχει το λόγο. Δεν έχουμε χρόνο πολύ, δεν θα σας επιβάλλω από όλου τους περιορισμούς, αλλά λογικά πλαίσια. Θα μιλήσω πολωνικά γιατί θα είναι πιο εύκολο για μένα. έχω τίποτα. Λοιπόν, πιστεύω ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε μια σύνοψη ε, απάντησης, μια συνοπτική μάλλον απάντηση. Ως προς την αιρεσιμότητα, ε, νομίζω ότι οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν περισσότερο στο μακροοικονομικό. Όσον αφορά τώρα τα, τα σχέδια υποδομών, τα, τα έργα υποδομών, θα ήθελα να πω ότι σύμφωνα με τις ε, ενώσεις εργοδοτών είναι απαραίτητο να, ε, να καλύπτονται ορισμένοι όροι. Δηλαδή, αν πρόκειται το χρήμα να δαπανηθεί αποτελεσματικά, οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, παραδείγματος χάρη θα πρέπει η υποστήριξη για τους ανέργους να είναι αποτελεσματική. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για να μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υλοποιήθηκε ο στόχος. Προϋποθέσεις λοιπόν, όρι, πλαίσιο, το οποίο συνοδεύει το έργο. Αυτό είναι απαραίτητο όσον αφορά το έργο το ίδιο, το σχέδιο. Πρέπει να πω ότι το σύστημα αξιολόγηση υπάρχει βεβαίως στο επίπεδο της συγχρηματοδότησης, τουλάχιστον στην Πολωνία, εξαρτάται από, το, από τα αποτελέσματα που θα επιτευθούν. Δηλαδή, αν συμφωνήσουμε ότι θα στοχεύσουμε σε ένα αριθμό συμμετεχών στο έργο και δεν εξασφαλιστεί ο αριθμός των συμμετεχόντων, τότε δι, ε, εισπράττονται λιγότερα κονδύλια. Δηλαδή υπάρχει μια αιρεσιμότητα, υπάρχουν προϋποθέσεις, αλλά είναι αρκετά απλουστευμένα. Δηλαδή πόσα χρήματα θα δεποτηθούν με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων. Αλλά δεν γίνεται μετά μια ανάλυση για να δούμε τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι μετά την κατάρτιση. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται κυρίως από τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της στήριξης. Δηλαδή από τον προσδιορισμό που γίνεται στην αρχή. Δεν μπορώ συνεπώς να σας δώσω απλή απάντηση αναρωτηθήκατε τι ευρύτητα πρέπει να έχει το Ταμείο. Μα αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Βεβαίως οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι είναι εκείνες οι οποίες επιτρέπουν στους ανθρώπους να βελτιώσουν την κατάστασή τους μακροπρόθεσμα. Διαφωνώ όμως με τις προτάσεις οι οποίες θέλουν την αντικατάσταση των κοινωνικών κονδυλίων των εθνικών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Θεωρώ ότι εδώ μιλάμε για μια αναπλήρωση πολύ απλή του εθνικού προϋπολογισμού και δεν αιτιολογεί την χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου. Συνεπώς και η ορατότητα, η δημοσιότητα του Ταμείου αποδυναμώνεται. Δεν ξέρω αν κατάλαβα πολύ καλά την τοποθέτηση των εργοδοτών και τους μηχανισμούς που χρηματοδοτούν τις αρχικές δραστηριότητες. Πρέπει να σας πω ότι πολλές χώρες είχαν ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Δηλαδή η βοήθεια η οποία δίνεται σε αυτό το αρχικό στάδιο είναι πολύ αποτελεσματική. Είναι ένα από τα εργαλεία τα πιο ε, ε, ευρεία χρήσεως. Δηλαδή, βοηθάει την εκκίνηση του επιχειρηματία. Θέλω να απαντήσω σε μία ερώτηση. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα. Τη δυνατότητα απορρόφησης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα ε, για το έκτο Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες πράγματι δεν ξέρουν πώς να, λειτουργήσουν, να χρησιμοποιήσουν μεγιστοποιώντας τα κονδύλια. Γενικά όμως η εικόνα είναι καλή. Δαπανώνται τα κονδύλια αρκετά γρήγορα, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος. Ε, πρέπει να αναρωτηθούμε αν οι, αυτοί που έπρεπε να ωφεληθούν ωφελούνται πράγματι. Ευχαριστώ. Και τώρα θα θα ήθελα να ζητήσω από τις άλλες κυρίες να αφήσουν τον κύριο Ρόιτερ να πάρει το λόγο γιατί έχει να πάει σε, μια συνάντηση. Αγγλικά ή γαλλικά θα μιλήσουμε όλοι γιατί σε λίγο θα χάσουμε και τους διερμηνείς στις 12.30. Έχουμε για, τις, για τα νέα επαγγέλματα και λοιπά με τρογγυλή τράπεζα σχετικά με τα ερωτήματα, να μην τα παριθμίσω όλα, αλλά να πω για ορισμένα από αυτά. Αυτό που ρωτήσατε εσείς ε, πώς εξελίσσονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας. Να δούμε ποιες είναι αυτές ε, σε σχέση με τις εργασίες που προτείνονται, τις θέσεις αυτές, είτε με εξωπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, κάτι άλλο και στις πολιτικές περί εκεί που υπάρχει κακός προσανατολισμός με κακές ιδέες, είναι το άμεσο και όχι το ε, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και υπάρχουν εξελίξεις στην αγορά εργασίας, υπάρχει το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο και σε τοπικό και περιφερειακό. Και επειδή πολύ τοπικό και περιφερειακό αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς ε, τι χρειαζόμαστε εταιρική σχέση. Και αυτοί που έδωσαν μια απόδειξη ήταν οι εταιρικέ σχέσει με του κοινωνικού εταίρου ε, και ανάμεσα στο δημόσιο και στι διάφορε ενώσει. Όπω σα είπα, εμεί παρεμβαίνουμε και σε ένα τομέα που είναι εκτό κυκλώματο ε, τα διάφορα άτομα και προσπαθούμε να τα φέρουμε μέσα στο κύκλωμα. Να δούμε λοιπόν, όχι να ανακαλύψουμε και πάλι τον τροχό, αλλά ένα μέρο είναι το δημόσιο, ένα άλλο από τους ε, εταίρους, ε, τους κοινωνικούς και άλλο από τις διάφορες ενώσεις και οργανώσεις ε, που προτείνουν αυτή την σωμάτωση ή που εργάζονται βάσει προσόντων. Και ακριβώς το πρόβλημα σήμερα δεν είναι ότι χρειάζονται νέες εταιρικές σχέσεις, αλλά σήμερα ποιο είναι το θέμα, ότι σε διάφορα κράτη-μέλη θα πρέπει να δούμε καθαρά ποια είναι αυτή η αρχή, γιατί σαν αποκλείονται, ξέρω το παράδειγμα της Ρουμανίας όπως και άλλων χωρών που άλλοι εκτός από τους κλασικούς ε, το δημόσιο και τις ενό κλπ. δεν συμφωνούν και επειδή υπάρχει κάτι μια σύγχυση ανάμεσα στα πόσα μέσα διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και άλλα μέσα για επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, ακριβώς εκεί παρουσιάζεται ένα πρόβλημα. Καταλήγω στο εξή. Πώ να δούμε, πώ να εκτιμήσουμε αν επιτυχάνουν αυτά τα μέσα, να δούμε πόσα άτομα βρίσκουν θέση και μάλιστα ποιοτικέ θέσει, εργασία ποιοτική και σταθερή. Και επίση, άλλο ένα, ο κοινωνικό παράγοντα ε, και στην στη Γαλλία κυρίω ε, από το 19 και μετά εργαστήκαν πας αυτό το πώ ε, από αυτή την ακινησία θα μετακινηθούν τα διάφορα άτομοι είναι κάτι που δεν μετρείται όμω αμέσω, ε, από τη στιγμή που θα βρουν δηλαδή μια θέση αλλά θα πρέπει να μετακινηθούν αυτά τα άτομα προ κάτι το σταθερό και μιλήσαμε για την Ευρώπη του 2020 όπω επίση και την πλατφόρμα κατά τη φτώχεια και κάπω αυτούς του ματωρισμού του χάνουμε από τον ορίζοντα πάνω σε αυτά και πράγματα που έχει έχετε ήδη ψηφίσει, αλλά βλέπουμε ότι προσέχουμε ιδιαίτερα μόνο την απασχόληση και μόνο την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, χωρίς να καταλαβαίνουμε πώς θα τους οδηγήσουμε προς την απασχόληση, τα προσόντα κλπ. Και αυτό είναι ένα μέλημα επίσης, να δούμε πώς θα δούμε καθαρά την ανάγκη που υπάρχει για την απαραίτητη επένδυση. Ευχαριστώ. Πολύ καλή στρογγυλή τράπεζα σας εύχομαι στην συμμετοχή σας. Θα συνεχίσουμε σύμφωνα με τη σειρά και... Ε, ναι, έχετε το λόγο. Πριν να φύγει ο κ. Ρόιτερ, καλό θα ήταν να ακούσει τη θέση της Νομοσπονδίας μας. Δεν πρόκειται εδώ για μάχη ανάμεσα σε εταίρους σε επίπεδο κοινωνικού ταμείου. Να μιλήσω τώρα, εντάξει σοβαρά. Δεν νομίζω ότι οι αγώνε μα είναι διαφορετική φύσεω. Σίγουρα με κυβερνητικέ οργανώσει και ευτυχώ ευτυχώ ασχολούνται με του πτωχούς επίσης όμως και συνδικαλιστικές οργανώσει, όχι όλε, βέβαια, που ασχολούνται με τους άνεργους, με τους πτωχούς και να πω από πλευρά μου, αυτό είναι το σύνθημα άλλωστε του Βελγίου, ώστε να φαίνεται καθαρά, η Ένωση φέρνει τη δύναμη. Έχουμε τον ίδιο αγώνα, τη διαμάχη για να ξεφύγουν από τη φτώχεια και μέσω μια εργασία. ξεφεύγει κανείς, ε, πετύχει, χαίνει ε, αξιόλογες συνθήκες, ε, ένα καλό επίπεδο. Κάτι που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης είναι ότι υπάρχουν φτωχές εργασίες, ας τις πούμε έτσι, και φτωχοί εργαζόμενοι και για να έχουμε ποιοτικέ θέσεις που να μην έτσι προσωρινές θέσεις εργασίας όπως συμβαίνει σε διάφορες χώρες. Και σίγουρα το κοινωνικό ταμείο αποτελεί το μέσο, το όργανο, το εργαλείο για να πετύχει κανείς το στόχο του, αλλά εμεί τι φοβόμαστε. Κοιτάζοντας ε, την στρατηγικές ε, προοπτικές του 2020 και τους στόχους ε, Κύριε Πρόεδρε, σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπω και τα διαρθρωτικά ταμεία τα υπόλοιπα, θα χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή αυτή τη στρατηγική του 2020. Όχι όμω με οποιοδήποτε τρόπο και ποια στρατηγική. Για μα ποιο είναι το σημαντικό, το ουσιαστικό. Αυτή η βάση αυτός ο πυλώνας ε, που είναι η ανάπτυξη που περιλαμβάνει όλους ε, θα πρέπει να αποτελεί τη βάση. Είναι βέβαια μια πρωτοβουλία για την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και δεύτερο αυτό το μέρος της αγώνα κατά της φτώχειας. Ε, βέβαια λαμβάντας υπόψη ότι αυτή η στόχη που έχει ψηφίσει το Συμβούλιο κατά 20 εκατομμύρια μείωση των πτωχών μέχρι το 2020 αυτό το φτωχό πληθυσμό 120 εκατομμύρια ακριβώς άτομα με την ευρωπαϊκή κρίση δυστυχώς Κάθε μέρα βλέπουμε την αύξηση αντίθετα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά λιμνάζουν, αλλά στην όλη συζήτηση και στη χρηματοδότηση πρόκειται για μια πρόκληση και να πούμε ότι ναι, αυτά θα πρέπει να συνδυάζονται, να συνδεδεμένα με τη στρατηγική του 2020, όπως επίσης και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη λήψη αποφάσεως, να δούμε ποια είναι αυτά τα στρατηγικά πλαίσια στον προσδιορισμό τους. Επίσης κάτι για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να μην αρκεστούμε μόνο στις κατευθυντέ γραμμές ε, με τις μέχρι τώρα γραμμές που υπάρχουν. Διαφορετικά ε, δεν θα μείνει τίποτα από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόληση ε, και μετά από τις αποφάσεις τελικά θα πρέπει να δούμε ποιο κοφή είναι αυτό που τα κάνει όλα και όχι στο Θα πρέπει να πούμε βέβαια, εμεί το λέμε, ναι, αυτέ είναι οι γραμμέ, βάση για την απασχόληση, αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε και τι προτεραιότητε, να τι επαναεπιβεβαιώσουμε, να υπάρξει μια, ασκηθεί μια ε, πολιτική πραγματικά και συμμετοχή κοινωνική ε, και επίση με στόχου που θα πρέπει να λάβουμε όπω ε, η ισότητα των φύλων από τη στιγμή την πρωτοβουλία αυτή που την εγκαταλείψαμε για τα φύλλα, τα ισότιμα, τι είδαμε. Ε, κανονικά θα έπρεπε να βλέπουμε ότι εγκαταλείφθηκε αυτή η θέση μεταξύ των κρατών και η εκτίμηση όλων αυτών ε, βλέπουμε μια πιστοχώρηση, πιστοδρόμηση και αυτά που σας λέω είναι πραγματικά σοβαρά. Στην περίπτωση αυτής της συζήτηση για τις συνθήκες, για τις προϋποθέσεις, εντάξει, ορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις θα πρέπει να γίνονται σεβαστές για την εφαρμογή των οδηγιών της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής και γιατί όχι και η ρύθμιση για την ισότητα των φύλων θα πρέπει να αποτελεί και μια προϋπόθεση για τα κονδύλια πώς θα δίδονται. Εντάξει, δεν έχουμε τα στοιχεία, θα πρέπει κανονικά να εμβαθύνουμε στην όλη συζήτηση και όλα αυτά τα συζητάμε με διάφορους που τα συζητάμε διάφορους που συναντάμε στους χώρους και βέβαια κάτι που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι παρουσιάζεται μια αυτονομία σχετικά με το ΦΕΝΤΕΡ, αλλά θα πρέπει να δούμε μια καλ... ένα καλύτερο συντονισμό με το ΦΕΝΤΕΡ, όπως επίσης και με τις υπόλοιπες ε, ευρωπαϊκές πολιτικές που ασκούνται, διαφορετικές άλλε γραμμές του προπολογισμού που συζητώνται και εδώ για το ΦΕΝΤΕΡ και για την εταιρική σχέση. Αυτό που ζητάμε, αυτό που απαιτούμε είναι μαζί με τις ε, ενό εργοδοτών αυτή η αρχή της εταιρικής σχέσης να συμπεριληφθεί στον κανονισμό του ΦΕΝΤΕΡ. Δεν υπάρχουν λοιπόν εκεί οι κοινωνικοί εταίροι, ούτε η τριμερής συμμετοχή κλπ. Ολοκληρώνω πολλά θα μπορούσα να πω ακόμα άλλα σχετικά με την εταιρική σχέση. Το ρωτήσατε αυτό, πάντως υπάρχει τρομερή απόσταση και μια κάποια χώρης, οπισθοδρόμηση ας πούμε και στις σκανδινεύικες χώρες. Ε, για ποιο λόγο η κατηγορία είναι ότι δεν υπάρχει πια κοινό ενδιαφέρον, απλά και μόνο είναι εδώ και εκεί που δίδονται, προσφέρονται κονδύλια και δεν ε, θα ενδιαφέρεται ίσως κανείς στο μέλλον. Αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί, επαναλαμβάνουμε. Και είπαμε σαν παράδειγμα όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, ολοκληρώσατε εδώ, γιατί έχω τρία λεπτά ακόμα για του δύο άλλου υπόλοιπου που θα πρέπει να λόγο. Με συγχωρείτε που σα αφαιρώ το λόγο, αλλά θα πρέπει να σεβαστούμε τον κόσμο εδώ. Βολεζίνσκι, λοιπόν, παρακαλώ, σύντομα, τηλεγραφικά. Ναι, η αγορά εργασία θα πρέπει να αποτελέσει το κύριο στοιχείο τη χρησιμοποίηση του κοινωνικού ταμείου σε κάθε διάσταση, συμπερίληψη κοινωνική, να δούμε νωρί-νωρί ποιε είναι οι ανάγκε δημιουργία θέσεων απασχόληση και μέσα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των βιοτεχνιών, ε, διαβίου κατάρτιση και αποτελεσματικό σύστημα και κατάρτιση, επαναλαμβάνομαι, από την αρχή, αρχή από τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό μέχρι παραπάνω και αυτονομία των δύο ε, οργάνων ε, ταμείων, αλλά ταυτόχρονα και συνεννόηση και συνεργασία. Ε, ναι. Έχουμε δύο προτεραιότητες που μας επιτρέπουν αρκετή ευκαμψία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι περιφέρειες και να δείξουν μέσω της διαφοροποίησης τους τις δυνατότητες τους. από το CRPM τώρα, επόμενος ομιλητής. Πολύ σύντομα και εγώ. Αν και είναι πολύ εκνευριστικό, διότι έχουμε πλούσια εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα και θα ήταν ενδιαφέρον να μπορέσουμε να τα συμμεριστούμε μαζί σας. Τέλος πάντων, πολύ σύντομα όσον αφορά την εποπτεία των αναγκών για την εργασία, για την απασχόληση, που είναι το πρώτο θέμα που θίξατε. Δηλαδή, πρέπει να φροντίσουμε να πάνε στην κατάρτιση αυτή που είναι η πιο απομακρυσμένη από τα απαιτούμενα προσόντα. Αυτό βεβαίως μπορεί να γίνει μόνο μαζί με τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και πρέπει να θεωρήσουμε την ενέργεια του, τις ενέργειες του ΕΚΤ μέσα στο πλαίσιο ενός τριγώνου. Δηλαδή έχουμε το κοινό, το πιο αποκομμένο θα έλεγα, την περιφέρεια και τις επιχειρήσεις τους κοινωνικούς εταίρους. Από την ώρα που έχουμε αυτό το τρίγωνο μπορούμε μαζί να ταυτοποιήσουμε τις αυριανές ανάγκες και ξέρουμε ότι τα επαγγέλματα τα αυριανά έχουν να κάνουν με την πράσινη ανάπτυξη. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο την κατεύθυνση του τεράστιου σκάφους της επαγγελματικής κατάρτισης και πρέπει να συνεργαστούμε με την περιφέρεια εγώ προέρχομαι από την Ακιτέν που είχαμε τεράστιες φυσικές καταστροφές στα δάση. Πρέπει συνεπώς τον πόρο, το ξύλο, τον φυσικό πόρο να τον αποκαταστήσουμε και συνεπώς αρχίζει μια νέα προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε τα, τα τεστραμμένα δέντρα κτλ. Όλα αυτά γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο. Τώρα όσον αφορά τη δεύτερη ευκαιρία, έφυγε ο μιλητής, αλλά αντί για δεύτερη ευκαιρία θα ήθελα να μιλήσουμε για νέα ευκαιρία. Πρέπει να ξεκινήσουμε όσο πιο νωρίς γίνεται. Να καταπολεμήσουμε παραδείγματο χάρη την εγκατάλειψη του σχολείου. Ε, είναι πολύ βασικό αυτό για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τους σωστούς για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες. Έχει αρχίσει αυτή η προσπάθεια. Είμαι δημοτική σύμβουλο σε μια, σε μια πόλη με 45% ε, ανεργία των νέων. Η εγκατάλειψη του σχολείου είναι ένα ουσιαστικό το στοιχείο. Πρέπει συνεπώς να παρακολουθήσουμε ολόκληρη την αλυσίδα. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε και απαντήσεις από το RCPM Αναφερθήκατε στις προτεραιότητες. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα ανανέωσης και καινοτομίας. Αυτό χρειάζεται το ευρύ κοινό περισσότερο και οι περιφέρειες επίσης. Η καινοτομία πρέπει να φεθεί πιο ελεύθερη, να πειραματιστεί, να δοκιμαστεί ό,τι είναι δυνατόν. Έχουμε περιθώρια διερεύνησης σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους. Αντιλαμβάνομαι πόσο ενδιαφέρεστε για αυτά τα θέματα και το έργο το οποίο πραγματοποιείται, αλλά έχει και αυτό το, και το Ευρωκοινοβούλιο τους κανόνες του. Ε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να καταλήξω σαν μόνιμη συγγήτρια. Έχετε ένα λεπτό και μόνο. Ωραία. Θα ήθελα να πω ότι αφού παρακολούθησα προσεκτικά τους κοινωνικούς εταίρους, η μεγάλη δυσκολία είναι να αλλάξουμε κλίμακα σκέψης. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε το μέλλον για τους, αυτούς που δεν έχουν απασχόληση, αλλά πρέπει ακόμη να μπούμε στη σημερινή πραγματικότητα. Πρέπει να τα κάνουμε τα δύο ταυτόχρονα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς σήμερα είχαμε λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα να ξανακούσουμε τους κοινωνικούς μας εταίρους, ώστε να έχουμε μία συζήτηση μέσα στο πλαίσιο της μόνιμης ομάδας εργασίας μεταξύ συνδικάτων και ε, Ευρωκοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Και εγώ, σαν πρόεδρος, θα ήθελα να σας προτείνω, αν υπάρχουν σημαντικά μηνύματα τα οποία θα θέλατε να μας δώσετε γραπτά,